liebe Kolleginnen, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, σα καλωσορίζω θερμά στη σημερινή συνεδρίαση τη Επιτροπή μα και επειδή δεν είχα παρευρεθεί κατά την πρώτη μα ε, συνεδρίαση, ε, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλου σα ε, ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτο. Νομίζω πω όλοι θα το χρειαστούμε. Τώρα να περάσω κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω πω μπορούμε να την εγκρίνουμε ω έχει με μία μικρή μεταβολή. Δηλαδή θα αλλάξουμε τη σειρά μεταξύ των σημείων 13 και 14 της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή θα εξετάσουμε το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης πριν από το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πλήρως γλωσσικό καθεστώς με την εξαίρεση των Μαλτέζικων. Ε, και μάλιστα είχα ακούσει κάποια στιγμή διερμηνία ματέζικα και είναι ενδιαφέρουσα γλώσσα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ούτε κροατικά ούτε ελληνικά. Τώρα, ε, θα γίνει μια αλλαγή, ε, γιατί η συνάδελφο είναι Σούμπα την 31η Ιανουαρίου α, δεν θα είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν γνωρίζουμε ποιος θα την διαδεχτεί ακόμα, δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάποιο όνομα. Από εκεί και μετά έχουμε μια ανοιχτή συνεδρίαση ε, των συντονιστών στις 26 Ιανουαρίου από τις 2 στις 3 ώρα το απόγευμα και ο Ιταλός ε, Υπουργό Οικονομικών, ο κ. αν θα παρευρεθεί. Μα θυμίσει με την παρουσία του και αποφασίσαμε να είναι ανοιχτή αυτή η συνεδρίαση γιατί θεωρούμε πω ε, αυτό το ζήτημα μια ευρωπαϊκή, ενό ευρωπαϊκού συστήματο ασφάλιση κατά τη ανεργία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήζει βέβαια μια ιδιαίτερα εντατική συζήτηση. Οπότε θα ήθελα να σα ε, καλέσω να παρευρεθείτε όλοι εκεί. Είπαμε ότι θα διαρκέσει μόνο μία ώρα σχετική ε, συνεδρίαση, δηλαδή από τις 2 στις 3 το απόγευμα, ελπίζω να παρευρεθείτε εκεί. Από εκεί και μετά θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας στην ε, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, η οποία ξεκινάει ή μάλλον θα λάβει η μαλλον θα λαβει χωρα 16 και 17 Φεβρουαρίου εδώ στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες δηλαδή την πρώτη ημέρα θα υπάρχει μία ολομέλεια και από εκεί και μετά οι διάφορες διακοινοβουλευτικές επιτροπές θα συνδυάσουν, η Apple, Econ και Budget, από τις 3 ε, έως τις 6, παράλληλα θα συνδυάσουν λοιπόν αυτές οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές και ε, τα σημεία της ημερήσιας διάταξης αφορούν ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και εμείς σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας ε, τι είναι το κοινωνικό τριπλό α, αυτό το τριπλό α στο κοινωνικό επίπεδο δηλαδή ένας πυλώνας για κοινωνικά δικαιώματα που περιλαμβάνει και το ζήτημα ε, δημιουργία ενός ε, μηχανισμού ε, ρύθμιστων των, τιμών, των μισθών συγγνώμη, και από εκεί και μετά οι επενδυτικές πολιτικές ό,τι αφορά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οπότε σας καλώ να σημειώσετε στα ημερολόγια σας αυτές τις δύο ημέρες 16 και 17 Φεβρουαρίου. Μετά περνάμε στο σημείο 5 το debriefing, δηλαδή την ενημέρωση με της Επιτροπής της, ε, ε, μάλλον μιας αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας ε, στον ΩΣΑ, στην, Επιτροπή, στην Υπηρεσία για την Εργασία. Δεν βλέπω αν είναι ο συνάδελφος εδώ για να μας κάνει αυτή την ενημέρωση. Όχι, βλέπω ο δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ο Σπάχ ήταν μαζί και εκείνος ήταν μέλος εκείνης της αντιπροσωπείας, αλλά δεν τον βλέπω εδώ, οπότε δεν νομίζω πως θα ακούσουμε τον debriefing σήμερα εδώ. Δεν θέλω δηλαδή να σας ε, αναγνώσω τη σχετική έκθεση της αντιπροσωπείας από το γραπτό κείμενο, οπότε εγώ από την πλευρά μου δεν έχω κάτι να προσθέσει, δηλαδή ενημέρωση σε ό,τι αφορά ε, το debriefing. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε σε μια από τις ε, της ε, διατάξεις των επόμενων συνεδριάσεων μας αυτό το ζήτημα και ένα ένα ακόμα ζήτημα βέβαια είναι η έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων 3 και 7 Δεκεμβρίου. Δηλαδή δεν έλαβα κάποιε προτάσει για την τροποποίηση των ε, πρακτικών, οπότε θεωρώ πω εγκρίνονται τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Καλώ ε, περνάμε λοιπόν στι ε, ψηφοφορίε. Έχουμε τρία στοιχεία επί των οποίων θα ψηφίσουμε. Καταρχήν, πρώτο σημείο, νέα εργαλεία δευτικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Όχι, έχει αποσυρθεί η τροπολογία 2. Α, όχι, κάνω λάθος λέει ο πρόεδρος, δεν έχει αποσυρθεί, οπότε σε ό,τι αφορά την τροπολογία 2 λοιπόν υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Συμβαστική β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τοπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αλλά θα ήθελα να το ελέγξουμε ελέγχουμε λοιπόν εγκρίνεται λοιπόν μετά 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε το συνόλου του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Έχετε ψηφίσει όλοι. Άρα λοιπόν πέρασε τη ψηφοφορία. 37 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Οπότε εγκρίνεται. Τα συγχαρητήριά μας λοιπόν στην Εσύτρια περνάμε στο επόμενο σημείο, απαλλαγή δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις διάφορες υπηρεσίες και έχουμε καταρχήν τον γενικό προϋπολογισμό, το οποίο θα ψηφίσουμε, δηλαδή το Discharge 2014 EU General Budget, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τοπολογία 1 λοιπόν υπέρ, κατά, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Καλώς. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Μετά έχουμε την συμβαστική τοπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τοπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Θα ήθελα να ελέγξουμε. 4 λοιπόν. Αν ψηφίσατε όλοι στο το πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στην 6 υπέρ, κατά. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώ, οπότε θα ελέγξουμε και τροπολογία 6 ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ. Πέραση τη ψηφοφορία λοιπόν και εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε λοιπόν την 9. Πέραση τη ψηφοφορία εγκρίνεται η τροπολογία. Θέλω να έρθετε λίγο πιο ενεργή, να σηκώνετε λίγο πιο ψηλά τα χέρια. Ε, ξέρω είναι Δευτέρα, αλλά σας παρακαλώ. Λοιπόν, 10 υπέρ. Α, όχι, είναι σε δύο κομμάτια. Λοιπόν, split vote ψηφίσουμε επί του πρώτου τμήματος λοιπόν, reminds that και ούτω καθεξής, υπέρ λοιπόν, κατά. Ευχαριστώ Ενρίκε, που σήκωσε ψηλά το χέρι. Απορρίπτεται λοιπόν το πρώτο τμήμα. Παίρναμε στο δεύτερο τμήμα, highlights once again και ούτω καθεξής, υπέρ. Α, όχι. Α, όχι, καταπίκτη, λέω, προς το δεύτερο τμήμα. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά έχουμε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 δεν υπάρχει πλέον άρα 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου της νομοδότησης ηλεκτρονικά μια ψηφίσατε όλοι πέραση ψηφοφορίας 32 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και 3 αποχές. Οπότε εγκρίνεται αυτή η γνωμοδότηση. Περνάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το πρώτο τμήμα εδώ δεν θα το, το μηδέν δηλαδή, είναι κάτι το τεχνικό, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε από αυτό, οπότε ψηφίσουμε από της 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε και πάλι επί του συνόλου ηλεκτρονικά εάν ψηφίσατε όλοι Πέραση ψηφοφορία. Έχουμε 34 ψήφου υπέρ και 8 κατά. πότε εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματική Κατάρτισης. Αλλαγή για το 2014. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ψήφι υπέρ. Α, μάλλον εγκρίνεται. Αυτομάτως 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Α, μου ζητάτε να, εξετάσ... να ελέγξουμε την 4. Καλώς ελέγχουμε λοιπόν τροπολογία 4 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Πέρασε λοιπόν τη ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αν θέλει κάποιο να ελέγξουμε, ελέγχουμε. 5 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και ψηφοφορία επί του συνόλου ηλεκτρονικά τώρα. Αν ψηφίσατε όλοι. Κλείνουμε λοιπόν και με αυτήν την ψηφοφορία. 32 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν εδώ τις επιδόσεις οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1. Εάν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Τέσσερα, τέσσερα διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 4 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Μετά, τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ α όχι Έχουν, έχει αποσυρθεί στο συγγνώμη είναι λίγο δύσκολο έτσι πρώτη μέρα για μένα και η 10 λοιπόν έχει αποσυρθεί οπότε περνάμε στην 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου ηλεκτρονικά. Εάν ψηφίσατε όλοι κλείνουμε την ψηφοφορία. 27 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτό το τμήμα. Περνάμε στο Δήμο Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πάλι απαλλαγή του 2014, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε για το σύνολο και πάλι εδώ τη γνωμοδοτηση ηλεκτρονικά Ευχαριστώ. Πέραση τη ψηφοφορία. 27 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Μετά περνάμε στο Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωση και Εργασία. Και πάλι 2014. Η 1 λοιπόν υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 6 ε, καταπίπτει, οπότε περνάμε στην τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε και πάλι για το σύνολο ηλεκτρονικά. Αν ψήφισαν όλοι. πέρα στις προφορίες, 32 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και πάλι. Τα συγχαρητήριά μας στον εισηγητή. So, dann kommen wir Περνάμε τώρα στην θέση της ε, Γιούτα Σάνρουκ όπου ακόμα δεν ήμουν σίγουρος αν, έπρεπε θα, ε, αν θα έπρεπε να αφήσουμε να γίνει μια ψηφοφορία. Ε, γιατί βλέπω πως και οι συζητητές δεν το έχουν λάβει ιδιαίτερα υπόψη τους. Το ζήτημα των φίλων. Εντάξει, αυτή είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, ή ε, τελικά μπορούν να κάνουν μόνοι τους δουλειά οι γυναίκες εδώ ή θέλουν τη βοήθειά μας. Τέλος πάντων, τροπολογία 1 υπέρ λοιπόν. Α, όχι 4 διορθώνουν πρώτος. Τροπολογία 4 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική M. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική E. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 με split vote εδώ ως τη ψήφο για το πρώτο λοιπόν τμήμα calls in the context of all measures υπέρ κατά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Εάν ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία, 25 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική π. Α, όχι, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 38 ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Ε, 4 υπέρ, 34 κατά, εντάξει. Λοιπόν, πει τώρα. Υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική AA υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 59 αν δεν απατώμε ναι 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 61 λέει ο πρόεδρος α όχι όχι άρα περνάμε σε συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε σε τροπολογία 71 με προφορική τροπολογία από τον ψυχητή, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται, 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, περνάμε στην συμβαστική U, υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται, συμβαστική τροπολογία W, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία MA Συμβαστική τροπολογία MA λοιπόν υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά Είμαστε λοιπόν MA. Αν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στη συμβαστική V. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική x υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 1. Είμαστε στα 40 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία A, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε επί του συνόλου της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά φυσικά. Εάν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία με 35 ψήφους υπέρ και 8 κατά και μηδενικές αποχές. Τα θερμά μας συγχαρητήρια για την και στον εισηγητή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις ε, ψηφοφορίες μας ε, για σήμερα. Περνάμε λοιπόν στα επόμενα τώρα σημεία της τη διαταξής μας και συγκεκριμένα στο 12, κοινωνικό dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη για Μπάλα είναι Και φυσικά του δίνουμε καταρχήν το λόγο. Παρακαλώ. Merci, Monsieur le, le Président. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι που ήρθατε σήμερα στη συνεδρίαση. Θέλω να σας παρουσιάσω αυτή τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας και θα ξεκινήσω περιγράφοντας το γενικότερο πλαίσιο. Όλοι μας γνωρίζουμε πως κάθε μέρα η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο εύθραυστη. Η μία κρίση ακολουθεί την άλλη. Από το 2008 οικονομική, γεωπολιτική, προσφυγικό, ε, περιβάλλον, καταλαβαίνουμε το γεγονός πως υπάρχει, υπάρχουν ερωτηματικά για το πόσο στέρεη είναι η σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και της ίδιας Ευρώπης. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και γιατί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και είναι ένα συνέστημα το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο. Καταρχήν συγκροτήθηκε η Ευρώπη για πάρα πολλούς λόγους βασιζόμενοι κυρίως στον οικονομικό πυλώνα και θα το περιγράψω πιο λεπτομερώς στην ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων, δημιουργώντας μια εσωτερική αγορά όπου τα εμπορεύματα και οι άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να μετακινούνται ελευθέρως. Αυτό οδήγησε και σε ένα πολιτικό οικοδόμημα ευρωπαϊκό το οποίο είναι πια πιο στεναρό παρόλο που σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι να υπάρχει μια πολύ βαθιά στρέβλωση μεταξύ αφενός της ε, εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής Ευρώπης αφετέρου. Γιατί οι οικονομικές ελευθερίες αυτή τη στιγμή εναρμονίζονται όλο και περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εσωτερική αγορά έχει ολοκληρωθεί στους περισσότερους κλάδους. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εκκρεμότητες, υπάρχει το κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας, αλλά για το κοινωνικό κομμάτι βρισκόμαστε ακόμα σε προϊστορικό στάδιο σε σχέση με την οικονομική Ευρώπη, γιατί τα κράτη διατηρούν όλα τα δικαιώματα στο στη χάραξη κοινωνικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων εθνών, μεταξύ των διαφόρων λαών, μεταξύ των ίδιων των μισθωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια θέμητη, έναν αθέμητο κοινωνικό ανταγωνισμό, αλλά αυτό ισχύει ακόμα και για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες, που σήμερα αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και που χρειάζεται να δώσουν τη μάχη με άνισα όπλα για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, για να επενδύσουν, για να καινοτομήσουν και τελικά δεν μπορούν να το κάνουν μια και χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μια κοινωνική, ε, ένα κοινωνικό ανταγωνισμό ε, ε, από που ξεκινά από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο με αποτέλεσμα να μην έχουν τα οικονομικά μέσα να καταφέρουν αυτά τα οποία επιθυμούν. Και πού μας έχει οδηγήσει αυτό σε μια εσωστρέφεια αλλά και σε μια περιχαράκωση των εργαζομένων στις χώρες με υψηλούς μισθούς ε, που απορρίπτουν τους εργαζόμενους που προέρχονται από πιο αδύναμες οικονομίες γιατί τους θεωρούν απειλή. Επίσης έχουμε ε, τις οικονομίες των κρατών που έχουν ε, χαμηλότερα οικονομικά πρότυπα που κλείνουν τις ε, αγορές τους και που δεν προσφέρουν μία προστιθέμενη αξία εμπορική αλλά απλώ προωθούν ε, φθηνότερο εργατικό δυναμικό το οποίο μειώνει την παραγωγικότητά τους και δεν ε, βοηθάνε ε, με τον τρόπο αυτό καθόλου την Ευρώπη. Άρα λοιπόν ο αθέμητος κοινωνικός ανταγωνισμός, το κοινωνικό dumping έχει αρκετές συνέπειες. Καταρχήν ε, κάτι το οποίο μπορεί να διακυβέσει την ίδια την εσωτερική αγορά, αυτή τη διάκριση μεταξύ εύρωστων και αδύναμων οικονομιών. Δεύτερον, ανταγωνισμός και οικονομία. Το κοινωνικό ντάμπινγκ επηρεάζει όλα, όλους τους ε, κανόνες και δημιουργεί αποπληθωριστικές τάσεις από τις οποίες κινδυνεύει η Ευρώπη σήμερα. Επίσης έχουμε κοινωνικά προβλήματα, μια και καταλαβαίνουμε πόσο πιο έφραυση έχουν γίνει και σε επίπεδο προστασίας που λαμβάνουν οι ε, εργαζόμενοι αλλά και σε επίπεδο απολαβών γενικότερα και όλα αυτά δεν οδηγούν σε μια ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Άλλωστε το λέει συχνά ο πρόεδρο Γιούνκερ, αν δεν έχουμε το τριπλό α σε κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απομακρυνθούν από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Νομίζω πως η απάντηση είναι αρκετά απλή, αλλά συνάμα και πάρα πολύ περίπλοκη. Περίπλοκη γιατί δεν έχουμε τις ίδιες παραδόσεις στα κράτη μας, περίπλοκη γιατί είναι διαφορετικό το επίπεδο πολιτικής ευαισθητοποίησης, γιατί ε, υπάρχουν ε, διαφορετικοί βαθμοί ε, συγκρότησης της εσωτερικής αγοράς στα κράτη μας και πιστεύω πως σήμερα εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα το οποίο έχει παρουσιαστεί μπροστά μας είμαστε σε θέση να το κάνουμε αρκεί και στο σχέδιο αυτό το οποίο που σας παρουσιάζω έχω ένα σχέδιο απλώς γνωμοδότησης, δεν είναι η τελική μορφή, είναι να μιλήσουμε στους ε, κλάδους οι οποίοι συχνά με το θέμα αυτό του κοινωνικού ντάμπινγκ, δηλαδή οικοδομή, κατασκευαστικός κλάδος, μεταφορές. Είναι δυστυχώς στην αιχμή του προβλήματος σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται ε, στην Ευρώπη, θαλάσσιες μεταφορές, η Ευρωπαίοι ναυτικοί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με ένα τρόπο που θα έπρεπε ε, να μας προκαλεί ντροπή. Νομίζω σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας ζουν σε συνθήκες ε, αδιανόητες, όπως επίσης στις ε, εναέριες συγκοινωνίες και μεταφορές που δεν υπάρχει προστασία των εργαζομένων, αλλά και στις οδικές μεταφορές όπου ξέρουμε ότι έχουμε κάποια πρόοδο, αλλά ακόμα έχουμε πολλές εκκρεμότητες με το καμποτάζ, ή και με την ε, κοινωνική εναρμόνιση των δικαιωμάτων των οδηγών, για παράδειγμα. Επίσης, έχουμε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Εδώ βλέπουμε πως ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα, βλέπουμε πως η Επίτροπος κυρία Τάισεν μας είπε πως, Τίσεν μας είπε πως χρειάζεται μια μεγάλη αναθεώρηση, αλλά και μια στοχευμένη παράλληλη αναθεώρηση για τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα σήμερα, μια και γνωρίζουμε πως υπάρχουν προβλήματα και μάλιστα τα προβλήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το έχω πει άλλωστε και στη γνωμοδότησή μου. Καταρχήν, έλεγχος. Γιατί βέβαια όταν η νομοθεσία υπάρχει θα πρέπει και να εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, θα πρέπει να προχωρήσουμε με απλά βήματα, δηλαδή να κάνουμε σημαντικές προσπάθειες, έτσι ώστε οι επιθεωρήσεις στον εργασιακό χώρο να ε, συσχετιστούν με τις προσπάθειες που κάνουμε με την νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη, χωρίς να έχουμε επιπλέον γραφειοκρατία. Πώς μπορούν να έχουμε ένα σώμα επιθεωρητών που να μην είναι πολύ άριθμο, αλλά να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό παρόλα αυτά. Για παράδειγμα, όπως έχουμε την Αμερικανική ε, φορεία και με χειρουργικό τρόπο να παρεμβαίνουν ως μυστέρι ε, σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα με αποτρεπτικό τρόπο για το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε και την ουσία της οδηγίας. Δηλαδή, και πάλι τίποτα δεν είναι απλό, το γνωρίζουμε. Ας ανοίξουμε το θέμα. Το βασικό στοιχείο είναι το εξή Γνωρίζουμε που συνήθως θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ένα ε, μισθό που θα είναι αντίστοιχος με αυτόν που θα ελάμβαναν, όχι σε μεικτά βέβαια, ε, στην ε, χώρα καταγωγής τους. Και εκεί ξεκινά ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει η διαφορά λοιπόν και σε επίπεδο κοινωνικών εισφορών επί του μισθού, γιατί ξέρετε πως είναι ο εργοδότης η εταιρεία η οποία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τις κοινωνικές εισφορές στον αποσπασμένο εργαζόμενο που θα είναι όμως οι κοινωνικές εισφορές της χώρας προέλευσης. Και εδώ έχουμε μια διαφορά οικονομική. Οπότε, τι θα κάνουμε, θα τις εξισώσουμε. Μα αυτό θα δημιουργήσει άλλες τρευλώσεις. Πρέπει σήμερα λοιπόν να ε, φέρουμε μια νέα ισορροπία στο σύστημα αυτό εάν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνισμό μεταξύ όσων προέρχονται από χώρες με ε, χαμηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και εργάζονται σε χώρες με υψηλό επίπεδο. Και θα το κλείσω κύριε Πρόεδρε λέγοντας πως το τρίτο σημείο είναι να σκεφτούμε το πώς μπορούμε να έχουμε μια συνολική κοινωνική σύγκληση. Το συζητάμε πάρα πολύ. Η Επίτροπο κυρία ο πρόεδρο Γιούγκερ, μιλάμε για το τριπλό α της κοινωνικής Ευρώπης που αποτελούν ε, τους πυλώνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρώπη το 2006. Έφτασε λοιπόν η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί και για το θέμα αυτό. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ε, ξεκινά μια σειρά από ερωτήματα τα οποία εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε και να πούμε απλά, καταρχήν υπάρχει το θέμα του ελάχιστου μισθού. Το να υπάρχει ο ίδιο ε, ένας ίδιος ελάχιστος μισθός για όλη την Ευρώπη δεν γίνεται. Θα πρέπει να εξαρτάται από ε, το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου οι εργαζόμενοι είναι ε, πολύ ε, ε, εξελιγμένη πολύ ε, ευέλικτη Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατόφλι. δεν είναι ελάχιστο μισθό σαν αυτό που θεσπίζει το κράτο, αλλά είναι οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι αποφασίζουν ποιο είναι το ελάχιστο κατόφλι μισθού. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα διάφορα στοιχεία μεταξύ μα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαζόμαστε για να στείλουμε ένα μήνυμα στον Ευρωπαίο εργαζόμενο. Όποιο και να είναι όποια και να τα πολιτικά μας πιστεύω, νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει βεβαίως η εσωτερική αγορά και θα πρέπει να προσέξουμε τις ε, ε, ενδεχόμενες ελλείψεις συμμετρίας που μπορεί να την θέσουν σε κίνδυνο. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η σχέση Ευρωπαίων με το οικοδόμημα αυτό είναι λόγοι που μας οδηγούν στο να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και το να τον το κοινωνικό ανταγωνισμό. Προφανώς, το να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, το να ακούσουμε τις δικές σας ιδέες και τις διαμάχες που θα έχουμε και που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε θα μας βοηθήσουν στην σχέδιο αυτογνωμοδότηση που θέλει να αποτελέσει απλώς μια αφετηρία για τη συζήτηση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ τον Κιγιάν ε, ε, <clears throat> θα ήθελα πολύ να αρχίσω να δίνω το λόγο σε όλους αλλά θα πρέπει καταρχήν να δώσουμε το λόγο στους κοιότητες συζητητές για το είπε ο κύριος Σουμπλέσκα παρακαλώ. Ο κύριος Κάζα. Δυστυχώς η Ντανούτα δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Και όταν ψηφίζουμε και έχουμε και ψηφοφορία στη Δευτέρα είναι κάπως πιο περίπλοκο. Θα σας μεταφέρω τις απόψεις στην Τανούτα για το θέμα πάντως. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλάς γιατί μας έκανε μία πρόταση ιδιαίτερα αναλυτική, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να διαμορφώσουμε την τελική θέση της Επιτροπής μας. Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το κοινωνικό dumping έχει συζητηθεί σε πολλές χώρες, όπως επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει νομική προσπάθεια ορισμού του κοινωνικού ντάμπινγκ. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν σε κάποια κοινά μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Να διευκρινίσω εδώ, λέει η Ντανούτα, ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι σκόπιμη κατάχρηση υπαρχουσών εθνικών και κοινοτικών ρυθμίσεων έτσι ώστε να αποκτήσει κανείς ένα ειδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη μείωση του κόστους της εργασίας και το μη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι' αυτό θα θέλαμε λοιπόν η έκθεση αυτή να έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, επιβολή, καλύτερη επιβολή ε, των ε, υπαρχουσών νομικών ρυθμίσεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Δεύτερον, ενίσχυση και αποτελεσματικότητα στη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές, όπως επίσης και πιο αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις επιθεωρήσεις εργασίας και τις υπηρεσίες ελέγχου. Τρίτον, ανείχνευση και κατάργηση των, στα παραθυράκια τα οποία μπορεί να υπάρχουν για την αποφυγή εφαρμογής του νόμου. Περιλαμβάνονται επίσης και για την απόσπαση των εργαζομένων συγκεκριμένες προτάσεις. Να θυμίσω ότι τα κράτη-μέλη στην παρούσα φάση εφαρμόζουν, μεταφέρουν στην εθνική νομική αρχιτεκτονική τους τα θέματα αυτά που επηρεάζουν το κοινωνικό ντάμπινγκ. Τον Ιούνιο του 2016 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, γι' αυτό και απαιτείται να υπάρξει γρήγορη εφαρμογή των ρυθμίσεων. Προτείνει επίσης ο εισηγητής στην περίπτωση των αποσπάσεων της αρχής της ε, ίσης αμοιβή για την ίση εργασία στο συγκεκριμένο τόπο εργασίας. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα, λέγει η Ντανούτα Χουμνέρ Και μια τέτοια λύση θα οδηγούσε σε μια περαιτέρω διάσπαση της εσωτερικής αγοράς, σε μια αύξηση της φαιάς περιοχής, σε περισσότερο κοινωνικό ντάμπινγκ και λιγότερη κοινωνική συνοχή. Η οδηγία του 96 για τις αποσπάσεις περιλαμβάνει συγκεκριμένε ρήτρε για να υποχρεώνονται οι εργοδότες να σέβονται ελάχιστα επίπεδα προστασίας. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ρήτρα. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να στρέψουμε ειδικά την προσωπή μας ε, στους, ε, στους ιδιαίτερα κινητικούς εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών. Απαιτούνται περαιτέρω ορισμοί και ενίσχυση και εφαρμογή των κανόνων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δικαιωμάτων τους. Για να βελτιωθεί επίσης η κοινωνική σύγκληση στην Ευρώπη θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο το σύστημα της ελάχιστης αμοιβή του ελάχιστου εθνικού μισθού σύμφωνα με τις δικές τους πρακτικές και την κοινωτική εμπειρία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους συνεισηγητές και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια θετική άποψη για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, Ντεβιτ Κάζα. Πράγματι, θα έχει πολλά να συζητήσει με την Τανούτα τώρα για την ίσια του Μακιντάρ. Uh, thank uh, Κυρία Μακιντάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο αυτό και να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Για τη δική μου ομάδα, και δεν σας εκπλήσω, η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι τα δύο στοιχεία κλειδιά. Και θα θέλαμε να υπογραμμιστεί αυτό και στην έκθεση. Οτιδήποτε ξεπερνά αυτές τις δύο αρχές για μας είναι προβληματικό. Θέλω να φανούμε λογικοί, θέλω να φανούμε ρεαλιστές και να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με τον τρόπο που τις επιτρέπουν οι συνθήκες. Πρέπει επίσης να αφήσουμε χώρο ελιγμών στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους εθνικές παραδόσεις και στο χώρο αυτό της απασχόλησης αλλά σε χώρους όπως η ασφάλεια. Τώρα, το πακέτο για την κινητικότητα γνωρίζουμε πως θα συμπεριλαμβάνει τρία σημαντικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να μην κάνουμε μία προσπάθεια μέσω αυτής της γνωμοδότησης να προκαταβάλουμε τα όσα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτάσεις οποίες ε, περιμένουμε το χρόνο, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερα να τηρήσουμε μια, σχέση, μια στάση αναμονής, να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν και να μην προσπαθήσουμε να τους προλάβουμε. Δεν πρέπει καταρχήν να αγνοήσουμε τις αναμενόμενες προτάσεις και θα πρέπει παράλληλα να λάβουμε υπόψη μας και αποφάσεις τις οποίες έχουμε λάβει στο παρελθόν. Να αναγνωρίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο αυτή την πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία, η οποία είναι μια πρόσφατη εξέλιξη και ο κύριος Περίνσκι ξέρω πως εργάστηκε σκληρά πάνω στο θέμα αυτό και να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν εκεί κάποιες διατάξεις ε, ισχύουν και να μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο ή κάτι που ξεπερνά κάτι το οποίο μόλις αποφασίστηκε. Με διακατέχουν σοβαρές ανησυχίες για την, με την αρχή αυτή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο και δεν πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα λύσει το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ με οποιοδήποτε τρόπο. Και να ανοίξω μια παρένθεση. Πολλές φορές αγνοούμε παντελώς ε, τις ε, συνέπειες τις οποίες εμείς δεν έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, αν μιλάμε για τέτοιου είδους ίση αμοιβή για τους εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται από φτωχότερε χώρες. Τι θα κάνουμε για τους εργαζόμενους που ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Έχω προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω στείλει συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο να εργαστούν στην Ουγγαρία. Αν λοιπόν μπορούσαν να τους ε, πληρώσα μόνο τα όσα την, την Ουγγρική αμοιβή, θα είχαν αρνηθεί να πάνε. Και αν η Ουγγρική εταιρεία έπρεπε να πληρώσει όλους τους εργαζομένους της ε, την ίδια αμοιβή που προσφέρουμε σε αυτούς τους συμβούλους που φεύγουν το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, δεν θα άντεχαν. Οπότε μην ξεχνάτε πως αυτή η αρχή μπορεί να εφαρμοστεί ε, και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν θέλω να προδικάσω τι θα συμβεί με την οδηγία περί απόσπασης ε, ή με την αναθεώρηση, εν περιπτώσει, αυτής, αλλά η συνάδελφος Ντανούτα, η οποία σήμερα δεν είναι εδώ, συμφωνεί μαζί μου στο ότι θα πρέπει η οδηγία επί, περί επιβολής να έχει το χρόνο να δράσει, γιατί θα προστατεύσει κάπως παραπάνω τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους, να δούμε τι θα βγει από την αξιολόγηση και πιστεύω πως οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτής της οδηγίας θα έχει αρνητικές συνέπειες γιατί θα δημιουργήσει αβεβαιότητες για την εφαρμογή της οδηγίας περί επιβολής. Ε, πιστεύω πως δεν θα πρέπει καθόλου να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Τώρα για το θέμα των μεταφορών. Ξέρουμε πως η Επιτροπή Τραν αυτή τη στιγμή έχει γνωμοδότηση ε, παρόμοια με αυτή τη δική μας επιτροπή. Άρα λοιπόν η Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να ασχολείται με θέματα που είναι ε, της δικής μας ε, ε, αρμοδιότητας το καμποτάζ, ε, για παράδειγμα, ή το handling, είναι θέματα τα οποία από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Τραν δεν μπορούμε να τους τα να τους αφαιρέσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε το θέμα των πλασματικών αυτοαπασχολούμενων. Εμείς είμαστε χώρες σε, σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν ε, αρκετά ευέλικτο, ευέλικτο ορισμό και ελεύθερη ε, ελεύθερες σχέσεις αγοράς που επιτρέπει ε, μεγαλύτερη συμμετοχή από ομάδες εργασιακές οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν αποκλειστεί από το χώρο της εργασίας. Για την ε, κοινωνική σύγκληση είναι σημαντικό όταν αναφερόμαστε στο θέμα αυτό να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο. Η δική μου ομάδα πιστεύει πως πρώτα απ' όλα σημαίνει μία αύξηση των βέλτιων πρακτικών, ε, το, του benchmarking, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να στοχεύσουν στους κλάδους στους οποίους χρειάζεται να αναλάβουν δράση και που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη που το χρειάζονται να βοηθηθούν. Δεν σημαίνει το, το κοινωνικό benchmarking περισσότερη νομοθεσία, και δεν υπάρχει η δυνατότητα ε, ε, να εφαρμόσουμε νομοθεσία η οποία θα ισχύει με ίδιο με παρόμοιο τρόπο για όλους. Θα κλείσω λέγοντας πως οτιδήποτε προτείνουμε θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία για, την καλύτερη, ε, για τις καλύτερες ρυθμίσεις, για το better regulation και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίηση κάνουμε να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Τώρα, με χαρά προσμένω στη συνεργασία με τον εισηγητή και ήδη ε, το ανακοινώνω πως θα καταθέσουμε τροπολογίες. So, für die Alde hätte jetzt das Wort Ματίνα Λαμπαγιώβα. Αλλά ε, δεν την βλέπω να είναι εδώ, οπότε Μαρίνα, παρακαλώ. Ναι, θα μιλήσω εκ μέρους της Ματίνα. Καταρχήν Ματίνα θα ήθελα να ευχαριστήσει τον συγητή για την πραγματικά περιεκτική δουλειά που έκανε σε σχέση με αυτό το ε, σχέδιο έκθεση και αναμένει βέβαια με ενδιαφέρον την εταιρική συνεργασία μέσα στι επόμενε εβδομάδε. Κατά την άποψή τη, λοιπόν, είναι καλά διατυπωμένο αυτό το σχέδιο σε ό,τι αφορά κάποια βασικά ζητήματα, αλλά έχει να κάνει κάποια σχόλια. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά ε, αυτήν την αρχή ε, τη ίση αμοιβή για την ίδια, ε, ίδια εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα και στο πλαίσιο των μισθολογικών διαφορών. Ε, σε ό,τι αφορά του απεσπασμένου εργαζόμενου και, τη, σύγκρισή του, αν θέλετε, με του φυστάμενου. Ε, δηλαδή στους τοπικούς εργαζόμενους, είχαμε την η υφιστάμενη οδηγία, η οποία βέβαια ενισχύθηκε και με την οδηγία εφαρμογής της πρώτης οδηγίας του 2014 ε, ε, και θα αρχίσει η εφαρμογή της τον Ιούνιο του 2016. Άρα λοιπόν η εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας, η εφαρμογή του 2014 θα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη φέτος ήδη ούτως ώστε να εφαρμοστεί σωστά στην πράξη. Ε, ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το πλαίσιο ε, είναι λοιπόν αυτή η οδηγία η εφαρμοστική και γι' αυτό θα πρέπει να περιληφθεί και στη δική μας έκθεση. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τους ίσους μισθούς για τους αποσπασμένους και τους τοπικούς εργαζόμενους για την ίδια εργασία θα πρέπει θεωρούμε να αναφέρεται μόνο ε, σε σχέση με τον ελάχιστο ε, μισθό ο οποίος έχει συμφωνηθεί στο επίπεδο συλλογικών συμβάσεων εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν διαφορές σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους, ε, ή θα πρέπει και να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις εκάστοτε επιχειρήσεις ή στον τύπο του κάθε εργαζόμενου γιατί δεν θα είναι δυνατό να επιτύχουμε ίδιε αμοιβέ παντού και δεν θα επιτρέψει βέβαια και δεν θα δώσει τη δυνατότητα στι επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται τους μισθού με τους εργαζόμενου. Μετά, δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνει συνάδελφος αφορά τον τομέα των μεταφορών σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Μεριζόμαστε λοιπόν ε, την ε, πρόταση του εισηγητή για τη δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μεταφορών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά και του κανόνε για τα καποτάζ. Ε, καλό θα ήταν να γίνουν τέτοιε αναφορέ όπω και αναφορέ στα μέτρα εθνικά τα οποία λαμβάνονται και τα οποία δημιουργούν νόμικη αβεβαιότητα και αμφίβολα μέτρα σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει για επιχειρήσεις τη αλλοδαπής οι οποίες δραστηριοποιούνται ε, στην ε, Γερμανία. Και ε, βέβαια το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστοί αντίστοιχοι κανόνες της Επιτροπής. Επίσης, συνάδελφο ζητάει από τον εισηγητή να διευκρινίσει λίγο τις προσθέσεις του σε ό,τι αφορά την παράγραφο 21, η οποία αναφέρει ότι η, οποία, ε, ότι η Επιτροπή, τα πλοία τα οποία μεταφέρουν αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν, έχουν σημαία κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ανήκουν σε ε, ε και φυλακή Επίσης, σε σχέση με το ίδιο κεφάλαιο, τι ακριβώς προσπαθεί ο εισηγητής στην παράγραφο 25, παράγραφος 4 ε, να ε, πει με τα wage flows, τα επίπεδα δηλαδή των ε, μισθών. Και αν θεωρεί δηλαδή ο εισηγητής ότι αυτά τα flows θα πρέπει να δημιουργηθούν και σε ποιο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 λοιπόν παράγραφος εδάφιο 4. Από εκεί και μετά ε, οι σχετικοί κανόνες είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας είτε μέσω εθνικής νομοθεσία αποτελούν αρμοδιότητε λοιπόν των κρατών μελών και όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το άρθρο 153 τη Ένωση, το μόνο που μπορεί να κάνει εδώ η Ένωση είναι να ενισχύσει και να υποστηρίξει τι δραστηριότητε των κρατών μελών. Και βέβαια, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών επιπέδων ε, του ακαθάριστου ε, ε, προϊόντο μεταξύ των ανατολικών και των υπολείπων κρατών μελών, είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να γίνει σεβαστή και αρχή τη επικορικότητα. Τέλο, θα ήθελε η συνάδελφο να ευχαριστήσει εκ των προτέρων ε, τον εισηγητή για τη λήψη υπόψη των σχολείων της και αναμένει βέβαια με ενδιαφέρον τη συνεργασία με τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις ε, για αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Μαριάν Χάκιν για την ΚΟΕ τώρα. Ο κ. Σελικιώτης δεν είναι εδώ δυστυχώς. Θα αναλάβει λοιπόν το λόγο εργοδιασμό του κάποιος. Κανένας λοιπόν συζητήσει για την ΚΟΕ. Πράσινη λοιπόν. Καλή μαντελή, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η Ευρώπη νομίζω ότι θα χαρακτηριστεί από το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ένα από τα βασικά θέματα, το οποίο θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της εντολής μας από εδώ και πέρα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα με το οποίο καλούμεθα να ασχοληθούμε. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο κύριος Μπάλας. Έχουμε μια σωστή βάση για συζήτηση. Το κοινωνικό ντάμπινγκ καταρχάς είναι θέμα ελέγχου. Η εφαρμογή της αρχικής και της δευτερεύουσας οδηγίας και πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε αν δεν υπάρχει έλεγχος. Ένα από τα κλειδιά λοιπόν της έκθεσης αυτής είναι το θέμα ακριβώς του ελέγχου. Και σαν συντονίστρια της Επιτροπής Μεταφορών ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε αυτή την εποχή στην Επιτροπή Μεταφορών και στα πλαίσια της οδηγίας ε, για τους αποσπασμένους γιατί πολύ συχνά ξεχνάμε το θέμα της υπεργολαβίας, σαν παράδειγμα, και το τι σημαίνει για τους εργαζομένους. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι δείκτες στην έκθεση αυτή, οι οποίοι πρέπει να μας απασχολήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Καταρχάς, ένα ευρωπαϊκό σώμα ελεγκτών. Αυτή είναι μια ιδέα την οποία προωθούμε εδώ και πολύ καιρό και η οποία δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει εφαρμοστεί γιατί απαιτείται και δεν υπάρχει θέληση συντονισμού και γενικά η απαιτούμενη βούληση θα έλεγα πολιτικά στα διάφορα κρατημέλη. Το δεύτερο θέμα, ο δεύτερος δείκτης είναι το θέμα της ελάχιστης αμοιβή του ελάχιστου μισθού. Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη θα καθορίσει, ότι αυτή θα καθορίσει ένα ποσό για όλες τις χώρες, αυτό προφανώς είναι λάθος και υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε κάθε χώρα να θεσμοθετήσει ένα υψηλό επίπεδο. Είναι βασικό αυτό, είναι ένα απαραίτητο βήμα και για τον εργαζόμενο, αλλά επίσης ε, είναι θεμελιώδες και για την ευρωπαϊκή, την κοινωνική Ευρώπη, την οποία όλοι θα έλεγα υποστηρίζουμε, αλλά την οποία δεν βλέπουμε να απογειώνεται. Το θέμα λοιπόν του κοινωνικού ντάμπινγκ εφαρμόζεται ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Είδαμε τι γινόταν και στο κτίριο εδώ, είπαμε επίσης τι γινόταν και στο θέμα της βιομηχανίας τροφίμων. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τον κύριο Μπαλάς που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε εκ νέου τον τομέα και να βοηθήσουμε τους εργαζομένους που πολύ συχνά καταδικάζονται από τον στρεβλό ανταγωνισμό που υφίστανται. Ευχαριστούμε την ε, Λάουρα για την FTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαλάς για την πρότασή του, την αρχική, είναι μια πρόταση εν πολλής μπορούμε να την δεχτούμε. Όπως υπογράμμισαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συγκεντρηθούμε στο συγκεκριμένο θέμα γιατί το κοινωνικό ντάμπινγκ δημιουργεί στην Ευρώπη συνθήκες ζωής ε, που βρίσκονται στο αντίθετο των προσδοκιών του Ευρωπαίου πολίτη. Επιβάλλεται λοιπόν προς εμάς τους νομοθέτες να λάβουμε τις σωστές και αποτελεσματικές αποφάσεις. Αυτό το οποίο επίσης με βρίσκει σύμφωνη είναι κάποιες σκέψεις ε, που ακούστηκαν για μια ευρύτερη συζήτηση. Μιλάμε για τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε στρεβλή. Ε, η εσωτερική αγορά πάρα πολλές φορές προκαλεί ανισότητες και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν το δούμε με μια κάποια προοπτική και αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη, όταν επιτέλους εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσουμε να δώσουμε στην Κίνα το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Γιατί πάρα πολύ συχνά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ανταγωνισμός καθίσταται στρεβλός και άδικος. Καταλάβετε τώρα τι θα συμβεί όταν θελήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση σε οικονομίες όπως της Κίνας, όπου επιτρέπουν τη στήριξη της βιομηχανικής τους δραστηριότητας μερικές φορές σε ύψος που ξεπερνάει το 50%. Λοιπόν όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερο θάρρος και να κατανοήσουμε τι είναι η Ευρώπη, πού θέλει να πάει η Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων σήμερα. Σημερίζομαι αυτά που είπαν οι προηγούμενοι σχετικά με τους τομείς οι οποίοι κατά πλειοψηφία εμπλέκονται και ε, έχουν χτυπηθεί από το κοινωνικό ντάμπινγκ και ιδιαίτερα οι μεταφορές. Εκεί όπου πράγματι επιβάλλεται η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας είναι ο τομέας αυτός και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό της υπηρεσίας και τις οδικές μεταφορές για τις οποίες μέχρι τώρα δεν προβλέπεται μια ειδική υπηρεσία και να ορίσουμε σωστά επίσης και τους κανόνες του καμποτάζ, γιατί εν πολλής το κοινωνικό ντάμπινγκ συμβαίνει, γιατί οι κανόνες του καμποτάζ δεν είναι επαρκείς και δεν δίνουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τους ελέγχους ε, για τους ελέγχους και για μια σωστή ε, μορφή ανταγωνισμού. Και το πιλωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ένα επιπλέον βήμα, ενώ θα ήταν απαραίτητο να ε, χρονομετρήσουμε τον χρόνο εργασίας, τον αριθμό των ταξιδιών και τον αριθμό των χιλιόμετρων τα οποία διανύονται. Σήμερα η έλλειψη επαρκών κανόνων του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές είναι κάτι το οποίο σαφώς και δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό dumping. Σαν Επιτροπή Απασχόλησης χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ελάχιστης αμοιβή που επέβαλε πολύ η Γερμανία και προς αυτοκινητιστές οι οποίοι απλά περνούσαν σε φάση διαμετακόμισης από την χώρα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θέσω, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τους αερομεταφορείς. Ζω στην Ιταλία και πάρα πολύ συχνά η απόκτηση από πλευράς μη κοινοτικών αεροπορικών επιχειρήσεων, των εθνικών σε εισαγωγικά ε, αεροπορικών επιχειρήσεων, δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού ντάμπινγκ. Ναι, δεν προσφέρουν υψηλότερες αμοιβέ, αλλά εν τω μεταξύ ουσιαστικά μειώνουν ή εκμηδενίζουν τις κοινωνικές εγγυήσεις τις οποίες προέβλεπαν οι συλλογικές εθνικές συμβάσεις. Συνεπώς λοιπόν τίθεται το θέμα του να προσπαθήσουμε να δούμε εμείς και τι μπορούμε να παραχωρήσουμε απέναντι σε μια προσωρινή φάση αύξησης των αμοιβών που δεν παρέχει όμως απαιτούμενες, τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Αυτό είναι προφανές στις αερομεταφορές. Δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, αλλά στη δική μου είναι ξεκάθαρο μέσω μόνο της αύξησης των αμοιβών δεν αυξάνει κανείς αυτόματα την ανταγωνιστικότητα και τις συνθήκες εργασίας. Έτσι αυξάνοντας απλά κάποιες αμοιβέ, μειώνουμε τις εγγυήσει για την εργασία και μειώνουμε και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είμαι λοιπόν στην διάθεσή σας για συνεργασία αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί τα περισσότερα από τα θέματα τα οποία κατέθεσε ο συνάδελφος ανήκουν είναι αλήθεια και στην δυνατότητα εξέτασής τους από την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Αλλά νομίζω ότι και μέσω αυτής της έκθεσης μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μπιτσότου τώρα για το Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Δόκτωρ Βέλμαλαν θα λάβει το λόγο για να σας δώσει την άποψή μας για την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η περιγραφή που έγινε ως, για τα όσα μπορούμε εμείς να προσάψουμε στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα με βρήκε πολύ σύμφωνη γιατί αυτή τη στιγμή καταλήγουμε σε κάποιες ε, καταστάσεις με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για όλα τα ευρωπαϊκά έθνη και πέραν του κοινωνικών θεμάτων και αντί να αντιμετωπίζουμε τα αίτια, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό της Ευρώπης σήμερα. Το κοινωνικό ντάμπινγκ και για τους μισθούς και για τις εισφορές ε, και για το περιβάλλον μας οδηγούν στα ίδια. Για το περιβάλλον δεν θα μιλήσω πολύ. Δεν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ορίζει το ίδιο το πρόβλημα, το οποίο ε, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από το μισθολογικό dumping. Κάθε κράτος μετά από 50 χρόνια Ευρώπης κάνει ό,τι θέλει. Μετά από εξωτερικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν διαμορφώσει τη ζωή μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Κάθε κράτος δίνει τους μισθούς που μπορεί, ανάλογα με το πόσο πλούσιο είναι κάθε στιγμή. Μετά από 50 χρόνια, και το διαπιστώνουμε σήμερα με την Ελλάδα, οι μισθοί, για παράδειγμα, σε κάποια κράτη καταρακώνονται. Σε άλλες χώρες που ανθίζει η οικονομία, ανθίζει γιατί ξεκίνησαν είτε από μια πολύ στερή βάση είτε γιατί κατάφεραν να ξεπεράσουν ή ε, να παραγωνίσουν το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό που θα επιδιώξουμε, που είναι ένα κοινωνικό σύστημα ε, με ισότητα, με δικαιοσύνη και με δικαιώματα, θα πρέπει να δίνουμε μισθούς οι οποίοι θα βασίζονται βέβαια στην ε, εργασία, αλλά θα λαμβάνουν υπόψη και κάποιες άλλες παραμέτρους. Έχουμε εδώ μία γνωμοδότηση η οποία πουθενά δεν αναφέρεται στο ύψος των κοινωνικών εισφορών, που όμως αποτελεί και τον πυρήνα του προβλήματος που έχουμε με τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν μια οδηγία η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία εμείς επιδιώκουμε, γιατί δημιουργεί μεγαλύτερες αδικίες Οι εταιρείε στη Γαλλία, για παράδειγμα, απευθύνονται για να βρουν ε, εργάτες ε, για γεωργικές εργασίες ε, σε εταιρείε ισπανικές οι οποίες τους φέρουν από τη Λατινική Αμερική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσοι είναι από χώρε που έχουν χαμηλούς μισθούς έχουν τη τάση να μετακινηθούν προς χώρες με ψηλότερους μισθούς. Αυτό δεν σημαίνει πως οι κοινωνικές εισφορές δεν θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι του μισθού τους. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να δώσω κάποιες συμβουλές στον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε ε, την προσπάθεια ευελιξίας, γιατί υπάρχει μια τεράστια διαφορά εδώ, ε, το οποίο προσπαθούμε εμείς να ε, γεφυρώσουμε. Και για το θέμα των κοινωνικών εισφορών να σας πω πως η διεθνή συνεργασία για την κοινωνική προστασία για όσους είναι, για παράδειγμα, από τη Γαλλία ξεκίνησαν το 1890 με την προστασία των ναυτικών. Και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε δεν πάνε όλα τόσα πίσω, αλλά υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης με ενεργό τρόπο, με μια κοινωνική προστασία για οποιονδήποτε μετακινείτε. Σημειώνω πως η Ευρώπη των Βρυξελών ε, κατέστρεψε τα πάντα και σήμερα θα πρέπει να οικοδομήσουμε από τη βάση, όχι βασιζόμενοι στα όσα προτείνετε εσείς, θα καταθέσουμε προτάσεις και τολμώ να ε, πιστέψω και να ελπίσω πώς θα τις ε, ακούσετε και θα τις διαβάσετε με προσοχή. Για την Επιτροπή ο κύριος Κλέμαν έχει το λόγο. Ή τουλάχιστον αυτό το όνομα έχω εδώ εγώ σημειωμένο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος από την Επιτροπή θα βάλει το λόγο. Όχι, Πρόεδρε, έχετε το σωστό όνομα. Θα κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει μια πρώτη ανάλυση αυτού του σχεδίου έκθεσης. Ε, διαπιστώνουμε όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των όσων θίγει εδώ. Ε, Περιλαμβάνονται τι μελλοντικέ προτάσει που θα κάνουμε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητα για του αποσπασμένου ε, εργαζόμενου ή και τι προτάσει που θα κάνουμε για τον συντονισμό τη κοινωνική ε, ασφάλιση. Επίσης θα δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στον πυλώνα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και εδώ λοιπόν θα υπάρξουν προτάσει από την πλευρά τη Επιτροπή και ίσω θα έπρεπε να αναφέρω και την ε, πλατφόρμα για της εργασία, εργασίας, γιατί βέβαια γίνεται και επανειλημμένα αναφορά στην αδήλωτη εργασία, στο σχέδιο. Η πλατφόρμα λοιπόν δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη λειτουργία της, οπότε αναμένουμε την επίσημη υιοθέτηση ε, της ε, πλατφόρμας αυτής, αλλά σύντομα, μετά δηλαδή από την επίσημη υιοθέτηση, θα ξεκινήσουν και τα διοικητικά βήματα τους ώστε να τεθεί πραγματικά σε λειτουργία η πλατφόρμα της αντιλωτής εργασίας. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η Ολλανδική Προεδρία θα διοργανώσει σε δύο εβδομάδες από τώρα μία διάσκεψη σε ό,τι αφορά την αξιοπρεπή εργασία όπου θα έλεγα πως το 1 τρίτο τουλάχιστον των ζητημάτων που έχετε θέσει μέσα στο σχέδιο θα συζητηθούν και εκεί, σε εκείνη τη διάσκεψη. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, έχω εδώ στη, στον κατάλογο των ομιλητών εννέα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα κλείσω λοιπόν τώρα τον κατάλογο των ομιλητών, οπότε δύο λεπτά θα έχει ο κάθε ένας από τους ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο. Άρα λοιπόν βλέπω μόνο κάποιες κρυμάτσες λέει ο πρόεδρος, αλλά όχι αντιρρήσεις επίσημες για αυτήν την πρόταση για τα δύο λεπτά λοιπόν. Οπότε, η Ελίζαβετ Μονσάντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για μια εξαιρετική έκθεση για όλους, για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Θα ήθελα όμως και στα πλαίσια της γενικότερης αντίληψης την οποία έχουμε για την κοινωνική Ευρώπη και για την στήριξη των λαών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, να θέσω ορισμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Μπαλάς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά. Θεωρώ ότι γύρω από την ε, αντιμετώπιση του θέματος δεν είμαι βέβαια ότι η ανάμιξη διαφόρων τομέων όπως ο ναυτιλιακός, ο αεροπορικός και ο παραποτάμιος είναι η σωστή αντιμετώπιση, γιατί οι τρεις αυτοί τομείς διαφέρουν μεταξύ τους πάρα πολύ. Και οι λύσεις οι οποίες, ε, τις οποίες καλούμεθα να βρούμε είναι λύσεις σε προβλήματα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Αγαπητέ για να προχωρήσουμε θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ανακατηγορία, τα μεν μετά τα δε. Αν τα αντιμετωπίσουμε με συνολικό, με σφαιρικό τρόπο, τότε φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε. Δεύτερο σημείο, πάνω στο οποίο θα ήθελα το να πάρω το λόγο είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Μετά την παρατήρηση την οποία έκανα στην πρώτη φάση, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω με την πρότασή σας. Θα πρέπει, πιστεύω, να βρούμε με τις υπάρχουσες υπηρεσίες να δώσουμε απαντήσεις πολύ πιο συγκεκριμένες. Δεν ξεπέρασα το δίλεπτο, Πρόεδρε. Πυρίνσκι. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι είναι μια σημαντική έκθεση και η πρόταση έχει διατυπωθεί σωστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι εννοούμε με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές. Η πρώτη είναι η κατάχρηση της ίδιας της εργασίας που μπορεί να καταλήξει και στην δραστική σκληρή εκμετάλλευση. Και το δεύτερο είναι οι αντικειμενικές διαφορές ανάμεσα στο ύψος των αμοιβών και στο ύψος επίσης των κοινωνικών ωφελημάτων. Νομίζω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα λοιπόν. Πρώτον, απαιτείται μια πιο αυστηρή εφαρμογή των ρυθμίσεων των εργασιακών έτσι ώστε να μην υπάρξει εκμετάλλευση. Να καταπολεμήσουμε λοιπόν τα άσχημα παραδείγματα και να δημιουργήσουμε σωστό ανταγωνισμό και το δεύτερο είναι ο κοινωνικός εναρμονισμός, η κοινωνική σύγκληση. Νομίζω ότι και τα δύο θέματα τα οποία τέθηκαν και το θέμα δηλαδή των κοινωνικών ωφελημάτων και το θέμα των αμοιβών δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα ρυθμιστεί προς τα κάτω, αλλά είναι κάτι το οποίο θα βλέπει προς τα ανώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Και εδώ η απουσία της ευθύνης αυτών οι οποίοι πληρώνουν και η απουσία των ενδιάμεσων, της αλυσίδας δηλαδή προμήθειας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Η πλατφόρμα σαν παράδειγμα είναι κάτι μέσω της οποίας μπορούμε να βρούμε αποτελέσματα καλύτερα. Ρέγνα. Ευχαριστώ. Εγώ θα συγχαρώ τον Γιώμ γιατί ε, έχει αναφερθεί σωστά σωστά μια σε ό,τι αφορά τις εταιρείε γραμματοκιποτίου, ε, τους ε, επισφαλείς ε, τομείς, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περιλαμβάνονται ήδη στο σχέδιο της έκθεσης. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω εδώ και το οποίο μάλλον και δεν έχει συμπεριλάβει εδώ ο Γιώμ είναι το ζήτημα των γυναικών γιατί βέβαια πολύ συχνά τυχάνουν εκμετάλλευση στις γυναίκες έσκεμένα. Ε, πάντως θα τεθεί με σίγουρα αυτό προς συζήτηση στο πλαίσιο της συζήτησης που θα κάνουμε για αυτό το, ε, σχέδιο Πάντω Πάντως ε, τίθεται εδώ ένα βασικό ερώτημα του γιατί δηλαδή ήθελαν οι λαοί της Ευρώπης να συνενωθούν για να υπάρχει και περισσότερη κοινωνική ασφάλεια. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για κοινωνική ασφάλεια δεν μπορεί να κάνουμε λόγο για τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν λαμβάνει χώρα εκμετάλλευση των ανθρώπων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η γενική τάση, η γενική εξέλιξη είναι ανωδική και όχι καθοδική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με την Εύελιν. Αναγκήρυκε. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, ε, σκέφτεσαι και αναφέρθηκε σε αυτό και τα πω και εγώ από την πλευρά της ε, δικής μας ε, της δικής μας ομάδας ε, εν συντομία σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το κοινωνικό triple A το triple α όχι, ε, έχεις προχωρήσει λίγο. Σε δύο ακόμα, θα πρέπει να περάσουμε δύο ακόμα σημεία της σε διάταξη για να φτάσουμε στο κοινωνικό τριπλό α. Κάνεις λάθος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, δράζομαι εδώ τις ευκαιρίες που μου δίνετε να μιλήσω την τρίτη μου γλώσσα τα Σουηδικά. Να πω λοιπόν ότι και εμεί ε, θεωρούμε από την πλευρά μα ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο στο πλαίσιο τη δική μα Επιτροπή, αλλά στο πλαίσιο του συνόλου του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιτρέψουμε την, ε, το να παραμείνει σε ύπαρξη αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε εμά ω Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Ήδη δηλαδή υπάρχει μια τάση η οποία ασκείται πάνω μα, υπάρχουν δηλαδή ε, και στο πλαίσιο της γενικότερης ε, του φαινομένου της μετανάστευσης και περισσότερες συγκρούσεις, δηλαδή βλέπουμε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους να είναι διατεθειμένοι υπό καταστροφικές συνθήκες να ε, προτείνουν ε, την εργασία τους, να εργαστούν δηλαδή, αρκεί ε, να είναι σε θέση να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν και εμείς με τη δική μας στάση μέχρι στιγμής ουσιαστικά τροφοδοτούμε αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ, το διαιωνίζουμε και κατά συνέπεια θεωρώ ότι πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ η εισηγητής. Ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω ή να τονίσω ιδιαίτερα και το οποίο θα αναφέρω και στις ε, γραπτέ μου προτάσεις τροπολογιών είναι η κοινωνική εταίρη. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Ναι, δίνεται ήδη έμφαση στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να επιταθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αναφέρομαι εδώ στους ε, κοινωνικού εταίρου τη αγορά εργασία. Δηλαδή από τη μία πλευρά επιχειρήσει, εργοδότε και από την άλλη πλευρά συνδικαλιστικέ οργανώσει. Ευχαριστώ, ο Μπάκμαν. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ε, μία συνάδελφος από τη Γαλλία αναφέρθηκε από την Front National ε, σε μια καρικατούρα των εισαγωγικών. Όχι, αυτό είναι ανοησία. Δηλαδή δεν μπορούμε να αμφισβητούμε εδώ τελικά την ευφυή, αν θέλετε, ή το δίκτυο νοημοσύνης της Επιτροπής μας. Εντάξει κάνουμε λόγο εδώ για ένα ζήτημα, προφανώ η γενική συζήτηση ε, αφορά, όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος μας ε, και ο κ. Ε, Γιούκερ, όχι μόνο στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για παράδειγμα στην Επιτροπή, αλλά αναφερόμαστε και στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε προτάσεις οι οποίε δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να τι εφαρμόσουν. Ε, συμφωνούμε με το γενικότερο σκεπτικό του σχεδίου. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν ε, οι κατάλληλε αμοιβέ ε, για την εργασία των ανθρώπων. Ναι, εντάξει, οι σημερινέ λύσει που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη δεν είναι σωστέ και πράγματι θα πρέπει να αναλάβουν αυξημένο εδώ ρόλο οι ε, οι κοινωνικοί εταίροι και φυσικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το επιχείρημα που μας λέει ότι όταν έχουμε μετανάστες οι οποίοι έρχονται στις χώρες μας δεν θα ισχύουν αυτοί οι κανόνες για αυτούς. Ε, είναι κάτι το εσφαλμένο. Επίσης, ε, στην ε, παράγραφο 18 ε, Γιώμα αναφέρεσε στο γεγονό ότι κάποιες συγκεκριμένε υπηρεσίες διοικητικές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά του, των εδαφών, δηλαδή στο πλαίσιο των μεταφορών, θα πρέπει να βελτιωθούν. Όμως, Γιώμ, με τι προσπάθειε που έχουμε κάνει, με τι διαδηλώσει που έγιναν στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, οδήγησαν σε πραγματικά αποτελέσματα. Είχαμε δηλαδή εκπροσώπου από τα ίδια τα κράτη-μέλη υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη σε αυτό το ε, τομέα και δεν υπάρχει ένας υπερβολικός ανταγωνισμός ο οποίος δεν δίνει καμία ευκαιρία στους εργαζόμενους. Άρα θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη εδώ. μια ακόμα σημαντική διάσταση, η υποστήριξη των ανέργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω πως δεν μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ακριβώς υπάρχουν πολύ μεγάλες ε, διαφορές απόψεων. Πάντως σε γενικέ γραμμές ναι, είναι σωστό το σκεπτικό. Δηλαδή δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την ύπαρξη κοινωνικού ντάμπινγκ, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να υπάρξει εδώ ε, μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα αν θέλετε προστασία αλλά ταυτόχρονα και αυξημένο ρόλο των ε, κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ. Ε, Άγνης έχει επιστρέψει οπότε θα της δώσουμε κατευθείαν τον λόγο. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά ήμασταν στην Επιτροπή Ίντα με τον Ολλανδό Υπουργό Εμπορίου, οπότε χρειάστηκε να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των δύο επιτροπών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία διαφορετικά σημεία. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Γκυγιόμ για την ε, έκθεση την οποία προετοίμασε. Πιστεύω πως έχει φτάσει στα χέρια μας την κατάλληλη στιγμή. Δεύτερον, θα προτιμούσα κατά πολύ αυτή να είναι η πρώτη μας απόκριση στο πακέτο για την κινητικότητα των εργαζομένων, δηλαδή να ήταν στο αρχικό σχέδιο που προτείναμε στις 9 Δεκεμβρίου, αλλά μια και δεν μπορεί πια να συμβεί αυτό, ας ετοιμάσουμε εδώ μια πολύ καλή έκθεση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί και η τρίτη μου πρόταση είναι η εξής. Ο πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει υπογραμμίσει πολλές φορές πως χρειάζεται ίση αμοιβή για ίση εργασία. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε εμείς. Εγώ είμαι οπαδός του Προέδρου Ιούνκερ όταν δίνει σημασία στο θέμα αυτό. Ξέρω πως δίνει ιδιαίτερη σημασία και η Ολλανδική Προεδρία Και αν τα πράγματα πάνε κατευχή και η διάσκεψη στο Άμστερνταμ καταφέρει να προωθήσει το τόσο σημαντικό αυτό θέμα, γιατί θα πρέπει να μας ξαναεμπιστευθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και νομίζω ότι για αυτούς η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια έκκληση έτσι ώστε να δείξουμε όλοι αλληλεγγύη είναι ένα θέμα αλληλεγγύης για το χώρο της εργασίας, δεν ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλο, αλλά αμοιβόμαστε ε, παρομοίως για παρόμοια εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά, κύριε Πρόεδρε. Μια κοινή γλώσσα του, του ε, εισηγητή μας, λέει ο κύριος Καλβέ Σαμβρόν, και όχι μόνο του Μολιέρου νομίζω ότι ακόμα ε, κανείς δεν έχει ε, περιγράψει με σαφήνεια τι είναι το κοινωνικό dumping. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Κανείς δεν ξέρει καν τι σημαίνει ίση εργασία. Και εδώ, εδώ προσθέτουμε και μία ακόμα συγκεκριμένη άποψη που είναι το τριπλό α. Ευτυχώς αυτά θα τα πούμε αργότερα. Αλλά αυτό το οποίο με έβαλε στον πειρασμό να ζητήσω το λόγο ήταν η αρχική εξαιρετική ε, τοποθέτηση του κυρίου Μπάλλας και έχω πολλά σημεία στα οποία συμφωνώ μαζί του, αλλά έχω και άλλα σημεία με τα οποία έχω αντιρρήσει. Βέβαια δεν είμαι πολύ δημοφιλή όταν τα λεφτά στην ομάδα μου, αλλά η κοινωνική Ευρώπη για μένα είναι απαραίτητη. Ε, και εκεί βασίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πάνω σε αυτήν θα ξαναχτιστεί. Για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα εντάξει, ε, αυτό δεν με κάνει δημοφιλή βέβαια, αλλά το καταλαβαίνω και υπάρχουν κάποια στοιχεία όπως για παράδειγμα αυτό που είχα στο δικό μου πρόγραμμα είναι το Σώμα Επιθεωρητών στην Ευρώπη ή εκείνη η παλιά νομοθετική πράξη την οποία είχαμε στα ναυπηγεία κάποτε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μόντι με τον κλάδο αυτό στην Ευρώπη τελικά τι έγινε. Επίσης υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνώ. Εμείς δεν θα δημιουργήσουμε την Ευρώπη παρά μόνο εάν εξασφαλίσουμε τρία ουσιαστικά σημεία. Κινητικότητα, καταρχήν. Άρα λοιπόν για την οδηγία για τις αποσπάσεις να είμαστε προσεκτικοί. Μέσω καλών προθέσεων ας μην επιτρέψουμε να εισέλθει και πάλι ο προστευτισμός στην Ευρώπη και ας μην αποτρέψουμε τους ε, εργαζόμενους ε, να ε, ανταγωνιστούν ένα στον άλλο σε επίπεδο μισθολογικό. Ίσως θα πρέπει να γίνουν πιο αντικονιστικοί οι μισθοί. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο μου. Και τι σημαίνει αυτό. Αν είμαστε ε, εναντίον της κινητικότητας και υπέρ του προστατευτισμού, αυτό βέβαια ε, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα είναι κακό για τις χώρες με χαμηλούς μισθούς, αλλά τελικά μεσοπρόθεσμα θα θίξει τον ανταγωνισμό των πιο πλούσιων χωρών. Άρα λοιπόν να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί κινητικότητα, ε, ελεύθερος ανταγωνισμός και όχι προστατευτισμός για να προχωρήσει η Ευρώπη. Ε, nein, ich sage da jetzt nichts dazu. Ε, später vielleicht. Όχι, δεν θα κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτό, ίσως αργότερα. Κύριος Ματέ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαν Ευρωπαίος πολίτης, χωρίς τη θέλησή μου, και χωρίς την θέληση των Γάλλων γιατί είδαμε πως αγνοήθηκε η άποψή του στο δημοψήφισμα του 2005. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μπαλάς, εξαιρετική έκθεση και η διαπίστωση που κάνει για τον ευρωσκεπτικισμό, για την πολιτική οικοδόμηση της Ευρώπης και για τις πολιτικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τι άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Ας θέσω λοιπόν στον κύριο Μπαλάς κάποιες ερωτήσεις. Αυτή η επιθυμία με το ζόρι οικοδόμησης της Ευρώπης. Μήπως θυμίζει το βάτραχο που θέλησε να γίνει μεγαλύτερος από το βόδι. Γιατί νομίζω ότι 6, 8, 10 χώρες εντάξει, αλλά 28 χώρες το να ολοκληρωθούν και να ενοποιηθούν οι συνέπειες είναι σοβαρές. Κύριε Μπαλάς, μήπως ήταν σκόπιμα όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες οικονομικές και βιομηχανικές ομάδες. Και τελευταία ερώτηση κύριε Μπαλάς παρά την καλή θέληση την οποία ίσως έχετε για την δημιουργία της κοινωνικής σύγκλησης με τους ελάχιστους μισθούς, μήπως πρέπει να φοβηθούμε ότι στο τέλος αντί να πάμε προς τα, πάμε, τα πάνω, μήπως στην ουσία μειώσουμε τις αμοιβέ των εργαζομένων και μήπως συστηματικά, με αργό αλλά συστηματικό και βέβαιο τρόπο, καταστήσουμε τους εργαζόμενους φτωχότερους. Runde jetzt der Kollege. τελευταίος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση σε όλους τους ε, συναδέλφους. Ε, η οποία είναι εξής. Έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό πρόβλημα Προφανώ δηλαδή το κοινωνικό τάμπινγκ, αλλά καταρχήν θα πρέπει να το ορίσουμε καλώ αυτό το πρόβλημα. Όπω είπε ήδη κάποιο σήμερα εδώ, δεν θέλουμε να έχουμε μια καθοδική, μια πιο προ τα κάτω σύγκληση, αλλά μια ανωδική προ τα πάνω ε, σύγκληση. Δηλαδή γίνεται λόγος ε, για ε, την ίδια αμοιβή, για την ίδια εργασία, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλαμπ των πλουσίων χωρών στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η πραγματικότητα δεν είναι τέτοια. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη ε, πλούσια και δεν είναι ίδια τα επίπεδα των μισθών στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς θα θέλαμε οι μισθοί της χώρε Ανατολικής Ευρώπης να αυξηθούν ή θα θέλαμε να ήταν, εν πάση περιπτώσει, υψηλότεροι, αλλά πρόκειται και για ζήτημα εδώ ανταγωνιστικότητας των οικονομιών. Και ακριβώ για αυτόν τον λόγο και οι χώρε Ανατολική Ευρώπη είναι πιο ανταγωνιστικέ σε σύγκριση με τις χώρες, τι δυτικέ χώρε σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία. Ε, εγώ γνωρίζω πολύ καλά και τη Γερμανία και την Πολωνία κύριε Πρόεδρε γιατί έχω ζήσει για πολύ καιρό και στις δύο αυτές χώρες. Η κατάσταση λοιπόν είναι η εξή. Ε, στην ε, Γερμανία είναι πάρα πολύ ακριβές οι ίσονος αν θέλετε οι μικρότερες ε, εμβέλειας υπηρεσίες στον χώρο των μεταφορών. Εξαιρετικά ακριβές λοιπόν στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά για παράδειγμα στην Πολωνία έχουμε για παράδειγμα το νοσοκομείο νοσοκομιακό προσωπικό. Ή και ο τομέας ε, της ε, φροντίδας ε, κατοίκων, οι σχετικές λοιπόν υπηρεσίες, πάρα πολύ ευθυνές και κατά συνέπεια μεγάλο μέρος αυτών των υπηρεσιών παρέχονται στη Γερμανία από εργαζόμενους της Πολωνίας χωρίς δηλαδή αυτές τις ε, υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την ε, ε, Πολωνία σε τόσο χαμηλές τιμές δεν θα είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σχετικοί κλάδοι στη Γερμανία οπότε ναι μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε λόγο για κοινωνικό dumping για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά είμαστε πιο ρεαλιστές δηλαδή η Σουηδία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χώρε όπου η σχετική προστασία είναι υψηλότατη, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρο, δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλά. γιατί δεν θα καταφέρει να δώσει τι απαντήσει. Αλλά βλέπω τον, τον παρακολουθούσα και είδα ότι σημείωσε και σημείωνε τακτικά τα πάντα εδώ. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι θα τα θέσει στο πλαίσιο της συζήτησης των σχεδόν εισηγητών. Απλά επιτρέψτε μου να κάνω ένα-δυο σχόλια σε ό,τι αφορά την ειδικότερα μια-δυο παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Καλό θα ήταν κάποιοι λοιπόν να εξετάσουν καλύτερα το σύστημα που ισχύει στη χώρα του σε ό,τι αφορά ακριβώ την συμφωνία, σε ό,τι αφορά του ε, μισθού και επίση ενδεχομένω θα μπορούσαν να ρίξουν ε, μια ματιά στι αρχέ τη πολιτική οικονομία, πρώτο εξάμεινο. Δηλαδή, ε, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά και προϊόντα και υπηρεσίε, δεν υπάρχει κανένα όφελο για καμία εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, σημαντικό αυτό εγώ εντάξει δεν είμαι ίδιος, απλά ε, δίνω ένα-δυο θυσμότα για σκέψη. Τώρα, περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης σε ό,τι αφορά δηλαδή το κοινωνικό τρίπλο α, social triple A, οι εισηγητέ συζήτησαν τον Οκτώβριο ε, και τον Δεκέμβριο και αποφάσισαν να τεθεί λοιπόν ως προφορική ερώτηση σε αυτό το ζήτημα, ως question, γιατί ε, στο πλαίσιο διαφόρων ομιλιών, για και από την πλευρά του Ιωσάν Κλον Γιούνκερ και από την πλευρά άλλων βέβαια μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε ακούσει επανειλημμένα να γίνεται λόγος για αυτό το κοινωνικό triple A, το τριπλό α, χωρίς όμως να μπορούμε να καταλάβουμε τελικά ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της έννοιας. Ζητήσαμε ε, ε, μία ε, τέτοια συνάντηση με την κυρία Τάις να πάρουμε κάποιες εξηγήσεις. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή η συνάντηση, οπότε αποφασίσαμε να υπάρξει ένα τέτοιο oral question, μια προφορική ερώτηση. Ε, προφανώς λοιπόν εγώ προεδρεύω εδώ, δεν έχω δηλαδή συντάξει αυτήν την ε, ε, ερώτηση, αυτό έχει γίνει από τη γραμματεία, αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ με το περιεχόμενο αυτής της ερώτησης. Επίσης, να πω ότι οι τροπολογίες σε ό,τι αφορά αυτά το, αυτήν την ε, προφορική ερώτηση μπορεί να γίνει μόνο από αυτούς που την υποστηρίζουν, δηλαδή ε, τους συντονιστές και να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 25 ε, γραμμές αυτή η προφορική ερώτηση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν χωράσει στο σχετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ως προς το περιεχόμενο, ούτω ώστε να φτάσουμε σε, ε, στο να περιορίσουμε το σχετικό κείμενο στις 25 ε, σειρές. Οπότε το τονίζω αυτό, ούτως ώστε να ληφθεί και στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Να είμαστε λοιπόν λίγο σύντομοι και εδώ στις παρεμβάσεις μας. Καταρχήν ήταν το λόγο ο κ. Ντέιβιτ Κάζα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σωστά ε, το είπε στην ε, ομιλή που έκανε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου δήλωσε ο πρόεδρος Γιονκέρ πως έχει αυτή τη φιλοδοξία να γίνουμε ένα τριπλό κοινωνικό α. Έκτοτε πολλά έχουν λεχθεί, αλλά έχουμε διάφορες ερμηνείες του τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φιλοδοξία. Θα συμφωνήσω μαζί σας θα έπρεπε και θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε ποιος θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη ιδέα ενό τριπλού κοινωνικού Α και ποια είναι τα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Μα έχετε κάνει πολλέ ερωτήσει για το τι ακριβώ είναι αυτό το τριπλό Α και έχουμε μία σειρά από κοινωνικού δείκτε ε, μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο που το περιγράφουν. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της νέας έννοιας. Για το περιεχόμενο της ίδιας της ερώτησης πιστεύω πως το κείμενο ναι, έχει ισορροπία, αλλά διαφωνώ με κάποιες προτάσεις σε αυτή τη φάση για το ποιοι δείκτες θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Ελπίζω βαθιά πως η τελευταία πρόταση θα διαγραφεί γιατί αν δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει, αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το τριπλό α, νομίζω πως θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζουμε σε ποιο κλάδος θα δραστηριοποιηθούμε. Λοιπόν, το τελευταίο θα ήθελα να διαγραφεί. Δεν με κλείσει αυτή η παρατήρηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε αυτό το ερώτημα στον κύριο Γιούνκερ ως προς το τι ακριβώς εννοεί με αυτό το τριπλό α, γιατί περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να λάβουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά αυτό το τρυπό α. Για μένα είναι σημαντικό να λάβουμε ε, μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ούτως ώστε μέσω ακριβώς αυτού του εργαλείου της προφορικής ε, ερώτησης να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο ε, Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ άλλωστε δεν έθεσε ε, προσυζήτηση ε, μόνο το ζήτημα του τριπλού α, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλειας και βέβαια η κοινωνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πάρα πολύ από πραγματικά ένα τρίπλο α, μια αριστεία στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε τις δικές μας προτάσεις από την πλευρά της δικής μας πολιτικής ομάδας. Πάντως σε κάθε περίπτωση ε, θέλουμε να λάβει χώρα αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ και γίνεται όχι στο παραπέντε ας το πω έτσι. Ευχαριστώ. Άννα και λέει ο Πρόεδρος. Αν θέλεις εδώ θα ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ερώτηση. Ναι, Πρόεδρε, ξεκινάμε μια ε, συζήτηση λοιπόν εδώ σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ένα τελείω ε, καινοτόμο ώρα, δηλαδή το, το τριπλό α, και αυτό βέβαια για το συμφέρον των πολιτών μα. Όμω θα πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι πρόκειται για μια ε, προφορική ερώτηση, άρα δεν έχουμε οριστική τοποθέτηση από τη δική μα πλευρά. Κάνουμε απλά ένα διερευνητικού τύπου ερώτημα. Και εκείνο που είναι σημαντικό στι συζητήσει που θα κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με του κοινωνικού εταίρου και άλλου φορεί, είναι να ε, διευκρινίσουμε το ποιες είναι απαιτήσει για να επιτευχθεί ένα τριπλό α, να ε, επιτρέψουμε το να λάβει χώρα ένας επικοδομικός διάλογος, αν τελικά έχουμε την ευκαιρία να τον διεξάγουμε. Ας ε, παραμένει λοιπόν εδώ εδώ αυτή η ερώτηση, πραγματικά ερώτηση, ας μην γίνει ένα ψεύδο ψήφισμα, ας μην εισάγουμε εδώ, αν μην το φουσκώσουμε με διάφορες απόψεις από δική μας πλευρά. Ας θέσουμε συγκεκριμένα το ερώτημα και ας ζητήσουμε από την Επιτροπή πείτε μας επιτέλους με βάση συγκεκριμένα δεδομένα τι ακριβώς εννοείται. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ναι. Ε, καλό θα είναι να ξαναδιαβάσουμε το κείμενο γιατί πραγματικά εδώ θα δείτε ότι μόνο ερωτήσεις περιλαμβάνει αυτό το κείμενο της προφορικής ερώτησης. Δεν έχει δηλαδή κάποιες τοποθετήσεις, δεν είναι ψεύδο ψήφισμα όπως είπατε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά, μια και εδώ δεν υπάρχει προτιμούμενη γλώσσα. Την πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης, μου φάνηκε πως είναι έτσι μια, ένα πυροτέχνημα του κυρίου Γιούνκερ, μια ευφυής αποστροφή. Και είπα μην του δώσουμε σημασία. Από τότε το έχω σκεφτεί πολύ. Και είχα και την ευκαιρία να συζητήσω με την Επίτροπη την κυρία Τίσεν, η οποία μου είπε πως όντως ήταν μια πετυχημένη έκφραση αλλά η οποία απλώς υποδεικνύει την δεδηλωμένη επιθυμία της Επιτροπής κτλ. Τώρα, συμφωνώ με τα όσα πιστεύετε και εσείς και η Επιτροπή μας και όσοι συνέταξαν το κείμενο, Λοιπόν, αν δεν θέλατε να γίνει φασαρία, ας μην μιλούσατε. Γιατί, εάν πραγματικά ξέφυγε προσπαθώντας να κάνει τον έξυπνο, να μας εξηγήσει. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνική Ευρώπη. Γιατί νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό. Άρα λοιπόν εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία, συμφωνώ μαζί της, συντάσσομαι, εξαιρετικές ερωτήσεις έτσι ώστε να έρθει αντιμέτωπη με τα όσα πρέπει να κάνει και τα καθήκοντά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως και πολύ σωστά εκφράσει ο κύριος Κάσα, όμως δεν είναι δίκαιο να βάλουμε και το τελευταίο εδάφιο. Εγώ συμφωνώ να χρειαστεί να αντικρίσει τις υποχρεώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ρωτήσουμε τι θα κάνει, τι σημαίνει, ποια είναι η έννοια, πώς το περιγράφει, τι θα είναι, θα είναι κάποιος οίκος αξιολόγηση για παράδειγμα, αλλά όχι να την προσανατολίσουμε εμείς την απάντηση που θέλουμε να ακούσουμε, να απαντήσουμε την ησυχία της και αν δεν μας αρέσει η απάντηση, ορίστε. Θα βάλουμε το νερό εμείς στα βλάκια για να πετύχουμε αυτή την ευέλικτη αγορά εργασίας κτλ. Και ό,τι θέλετε. Πρώτα να μας απαντήσει και μετά εμείς να αντιδράσουμε. Εγώ ποτέ, ποτέ θα δεν θα προσπαθούσα να προσανατολίσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομήνης και της τεράστιας ανεργίας που έχουμε σε κάποιες περιοχές. Μα με συγχωρείτε, για να είμαστε τριπλό α θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Και αυτό υπάρχει στο τελευταίο εδάφιο. Γι' αυτό, όπως και ο κύριος Κάσα, έτσι και εγώ προτείνω και θα προτείνω στην ομάδα μου. Και είναι σίγουρα εξαιρετική η σύνταξη, αλλά να βάλουμε τελεία και παύλα στο πρώτο τελευταίο εδάφιο. Και α απαντήσει ελεύθερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Bis zu dem Aber war ich schon richtig überrascht, Enrique. Ε, εξέπληξε με αυτό που σαν και πραγματικά. Τώρα, η Γκάμπη σήμερα για την Γκουε δεν την βλέπω όμω ε, εδώ στην αίθουσα, δεν ξέρω αν ε, αναλάβει κάποιος ο σκιώτης ο αγωγό τη Γκάμπη. Εάν όχι, το μας μέσα δεξιά του πράσινου λοιπόν. Νίχτ. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, ήταν η Τζιά; αλλά ούτε αυτή η συνάδελφο είναι εδώ για το ΙΕΝΑΦ, Ντομίνικ Ματά. Merci, Président. Relever le pilier social au même Λοιπόν, ο κοινωνικό πυλώνα, το να τον βάλουμε στο ίδιο επίπεδο με τον οικονομικό πυλώνα, νομίζω ότι είναι η έμονη ιδέα της Επιτροπή. Η στήριξη της κοινωνική Ευρώπη θα χρυσώσει εκ νέου την εικόνα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, ιδιαίτερα στα μάτια των ευρωσκεπτικιστών. Όμως, το άλοθη αυτό της πρόσδοσης κοινωνικού περιεχομένου στα ευρωπαϊκά προγράμματα θα επιβάλλει στα κράτη-μέλη μια ολόκληρη σειρά διαφθρωτικών αλλαγών για να σωθεί η Ευρωζώνη η οποία υπονομεύεται από μια πολύ διστακτική ανάκαμψη και από μια κοινωνική Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Η, η ανύψωση συγγνώμη, των κοινωνικών επιπέδων προστασίας θα δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά εργασίας. Το κράτος δικαίου έχει καταπονηθεί από τις δραστικές μειώσεις οι οποίες θα ανανεούνται αναεξαμηνιαία βάση εδώ και χρόνια. Συνεπώς λοιπόν η ανάπτυξη είναι δύσκολο να συνδυαστεί με πολιτικές υπέρ της εργασίας περισσότερο αποδοτικές από τις σημερινές. Άρα λοιπόν, ε, συν, συν σχολιαστές αν θέλετε, ολοκλήρωσαν. Ε, 5 Φεβρουαρίου λοιπόν το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών και συνέχεια θα γίνει ψηφοφορία. Επενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι μόνο οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων δικαιούνται να υποβάλουν τροπολογίες και επανθυμίζω επίσης ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τις κολπές σειρές σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διατύπωση του ερωτήματος και αυτό το λέω έτσι για να μην χρειαστεί τώρα να αρχίσουμε εδώ να κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις ε, για το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο τελικά δεν θα χωράει ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αλλά βλέπω ο κύριος ε, Κάσας θα το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, είχαμε εμάς την Άλντι και την ΕΣΥΑΡ που σας ζήτησαν να διαγραφεί σχετική παράγραφος και δεν ζητήσαμε να αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη παράγραφο αλλά να διαγραφεί απλώς. Ναι, ε, αλλά μιλάμε ότι κάποιος ε, άλλος από τους υπόλοιπους συν ε, εισηγητές αυτής της ε, πρότασης να έχει άλλη άποψη, να θέλει για παράδειγμα αυτή η παράγραφος να αντικατασταθεί με μια άλλη διατύπωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια σχετική πρόταση τροπολογία και από εκεί και μετά να συμφωνήσετε και να ψηφίσουμε τελικά. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια διατύπωση στην οποία, στην οποία θα συμφωνούμε όλοι μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε. Κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, δηλαδή και άκουσα την πρόταση που έγινε για τη διαγραφή αυτή τη τελευταία παραγράφου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την ε, θέση των υπολείπων πολιτικών ομάδων. Περνάμε λοιπόν ε, στο επόμενο σημείο τη διάταξη, δηλαδή το 13 το οποίο είπαμε ότι θα το διαθέσουμε ε, για λίγο πιο μετά. Φτώχεια, μια προοπτική με γνώμονα το φίλο. Λοιπόν, Λεν είναι συντάκτρια. Η αρμόδια βέβαια επιτροπή είναι η ΦΕΜ και εμείς ε, κάνουμε τη δική μας συνεισφορά σε ό,τι αφορά, δηλαδή τη δική μας γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την ένταση. Οπότε δίνουμε το λόγο κατευθείαν στην συντάκτρια της γνωμοδότησης κυρία Μπόιλεν. Ευχαριστώ πολύ το σχέδιο γνωμοδότηση είναι να αντιμετωπίσει αρκετούς παράγοντες που οδηγούν στην ε, μεγαλύτερη ε, φτώχεια των γυναικών ε, πληθυσμιακά στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει και πως είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που έχουν ε, μονογονεϊκές οικογένειες, όπως επίσης το γεγονός πως δεν μπαίνουν τόσο εύκολα στην αγορά εργασίας γιατί δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες δομές φροντίδας για τα παιδιά. Εγώ καλωσορίζω τους ε, σκιώδεις σε αυτή την γνωμοδότηση για να φτιάξουμε μαζί τις λύσεις για το πρόβλημα αυτό στα πλαίσια της δικής μας αρμοδιότητας. Το χρονοδιάγραμμα είναι μάλλον σύντομο. Στις βασικές ε, παραγράφους προσπάθησα να καλύψω όλα τα θέματα και χαίρομαι που η Επιτροπή ΦΑΜ έχει ε, καλύψει το θέμα ε, της διαφοράς της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι στο 33% αυτή τη στιγμή έχουμε την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση ως γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που ζητά να εξαλειφθούν οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών. Η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πραγματογνωμοσύνη της για να κάνει μια συλλογική απογραφή του τι χρειάζεται ακριβώς για να κλείσει αυτή η ψαλίδα και ποια είναι τα μέτρα τα οποία λήφθησαν ήδη από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κρίνονται πετυχημένα και να εντοπίσουμε γιατί κάποια μέτρα απέτυχαν και πού. Για να αλλάξουμε το βάρος απόδειξης θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που μας υποδεικνύουν τα στοιχεία ότι Δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στα μυθολογικά συστήματα, κατηγορηποίηση ουδέτερος προς το φύλλο και επίσης πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ε, γυναικών ε, ε, σε ανώτατο στελεχειακό δυναμικό. Επίσης, ε, δομές φροντίδας για τα παιδιά, γονική άδεια, οι επιπτώσεις αυτών συζητιούνται σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης που έχουμε και μετά την απόσυρση της οδηγίας για την γονική άδεια ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτασε η ώρα εμείς να επιμείνουμε πως θα πρέπει με μια νέα νομοθεσία να καλύψουμε τις βασικές ε, κατηγορίες αδικών που είναι η γονική, για παράδειγμα, η μητρική, η πατρική κτλ. έτσι ώστε να μπορούν να είναι εξίσου στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και να υπάρχει ε, άφθονη προσφορά ε, βρεφονιπιακών σταθμών που να καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες. Κατά τη γνώμη μου και έχω πολύ λίγο χρόνο σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στην αύξηση του επίπεδου διαβίωσης, για παράδειγμα, στη μείωση της προσωρινής ή επισφαλούς εργασίας που οδηγεί σε φτωχοποίηση των γυναικών και επίσης να ε, προσφέρονται και ε, μισθοδοτούμενη άδεια για όσους έχουν αντιμετωπίσει ενδοοικογενειακή βία. Θα ήθελα λοιπόν στη γνωμοδότηση αυτή να τονίσω πως το να κλείσουμε την ψαλίδα, τη μισθολογική ψαλίδα δεν θα λύσει το πρόβλημα των γυναικών που ζουν στη φτώχεια. Θα προσφέρει όμως προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να έχουμε και κάποια επιπλέον μέτρα στήριξη στη γνωμοδότησή μας γιατί ξέρουμε πως ε, έχουν ε, δυσανάλογα πληγή από τη λιτότητα οι γυναίκες, κυρίως λόγω περικοπών ε, στο σύστημα προνοιακών επιδομάτων. Και έτσι θα πρέπει ε, να συνδεθεί ο τρόπος που θα αυξηθεί το ελάχιστο μισθό, πώς θα συνδεθεί η παραγωγικότητα με τη μισθοδοσία και πώς θα στηριχθούν οι συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις. Για όσους είναι χαμηλόμισθοι ή λαμβάνουν ε, είναι χαμηλό μέσο μισθή μάλλον, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε εμείς να προωθήσουμε κάποιες διατάξεις που θα τους στηρίξουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για κάποια θέματα που πρέπει εκεί να απαντηθούν. Για την επισφαλή εργασία, Εμεί στη γνωμοδότησή μα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πραγματογνωμοσύνη που έχουμε και τι επιπτώσει που έχει στι γυναίκε και η δική μου ομάδα πιστεύει πω το γεγονό πω έχει αυξηθεί αυτή η προσφορά αυτή τη εργασία, η οποία είναι επισφαλή, είναι προσωρινή, είναι κακοπληρωμένη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο χάραξη πολιτική. γιατί δυσανάλογα και πολλέ φορέ και ε, θελούσια υποχρεούνται σε τέτοιου είδου εργασίε, σε εργασία οι γυναίκε θα πρέπει εμείς να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση για να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό. Μπορούν να το κάνουν μέσω της εφαρμογής ε, των συστάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, όπως επίσης και μειώνοντας τις περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως επίσης και μείωση ε, του χρόνου ε, αυτών των συμβάσουν περιορισμένη διάρκεια, έτσι ώστε αυτέ να οδηγούν σε μια μόνιμη θέση εργασία. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και να αναγνωρίσουμε την πίεση που, ε, ε, που, από την οποία υποφέρουν οι γυναίκε που είναι και θύματα ενδοοικογενειακή βίας και το γεγονό πω δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία. Μια οικονομική ανεξαρτησία που πλαισιώνει τη δυνατότητα που έχουν να ξεφύγουν από τέτοιου είδους βίες καταστάσεις. Επίσης, οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν το δικαίωμα σε μισθοδοτούμενη άδεια πολλές φορές κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Ε, υπολογίστηκε το ποσοστό των γυναικών που έχασαν τη δουλειά τους στην Ισλανδία λόγω οικογενειακής βίας και βεβαίω οι γυναίκε αυτέ κινδυνεύουν περισσότερο και από τη φτώχεια. Σε κάποιε πολιτείε των ΗΠΑ, όπω η Ουάσιγκτον, οι εργαζόμενε οι οποίε αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν άδεια είτε για να παραστούν στο δικαστήριο είτε για ιατρικά ραντεβού. Αυτή η εναλλακτική υπάρχει και στην Αυστραλία, όπου ε, αποτελεί και τμήμα των συλλογικών συμφωνιών και ε, σύντομα θα αποτελέσει και συνταγματικό δικαίωμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να αποτελέσει κομμάτι του θεματολογίου μας. Είναι ένα σχέδιο πολύτιμο, όχι μόνο της Επιτροπής ΦΑΜ ή της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά του Κοινοβουλίου ε, ολοκλήρου του Κοινοβουλίου. Στο συμπέρασμα να σας πω πως μπορούμε να μειώσουμε ε, τη φτώχεια στις γυναίκες με πολλούς τρόπους και εγώ στηρίζω πολύ στεναρά την γνωμοδότηση ΦΑΜ για το θέμα που συζητάμε σήμερα και πιστεύω πως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πραγματογνωμοσύνη για θέματα που άπτονται της απασχόλησης και τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την ε, γενική αυτόχεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την Επιτροπή ΦΑΜ και θα χαρώ να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές και στα θέματα στα οποία έθιξα, αλλά και στα θέματα τα οποία οι ίδιοι θα κρίνουν πως θα πρέπει να συζητήσουμε στα πλαίσια της γνωμοδότησής μας. Ευχαριστούμε, Ελένη. Τώρα οι σκιώδεις εισηγητές έχουν το λόγο. Η Ρωμάνα Τόμς, λοιπόν, για το Βέλγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι φτώχεια αποτελεί ένα όλο ένα και πιο σημαντικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουμε όλο ένα και περισσότερους πολίτες μας ε, βρίσκονται σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ε, φτώχειας. Έτσι λοιπόν γίνεται ακόμα πιο σημαντικό να ληφθούν μέτρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Μπόλεμ που προετοίμασε αυτή την ε, γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής μας ε, αποτελεί μια πολύ καλή βάση. Είναι ναι μεν σύντομο το κείμενο της γνωμοδότησης αλλά παρόλα αυτά είμαι ε, βέβαιο ότι θα δώσει το έναυσμα για εκτεταμένες συζητήσεις. Και βέβαια θα υποβάλω κι εγώ μια-δυο τροπολογίες. Ένα ζήτημα τώρα το οποίο θα ήθελα να θέσω πιο συγκεκριμένα είναι το ζήτημα που αναφέρεται δηλαδή το δικαίωμα του να λάβει κανείς άδεια μεταποδοχών σε περίπτωση ε, βίας ε, οικογενειακής. Ε, πράγματι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή για οικογενειακή βία, οπότε από την άλλη όμως πλευρά δεν ξέρουμε κατά πόσο μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει λύση, αλλά σίγουρα θα κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις για αυτό το θέμα. Μαρία Αρένα τώρα έχει το λόγο. Merci Σας ευχαριστώ. Θα πάρω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας Μπλινκεβιτσίουτε που δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα και στην Επιτροπή Γυναικών είμαι και εγώ υπεύθυνη για την έκθεση αυτή κάτι το οποίο συνδέει αν θέλετε την φτώχεια από τη μία με με κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Όταν βάζουμε τα γυαλιά και βλέπουμε σαν γυναίκα, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες στίγονται περισσότερο στην Ευρώπη, είτε οι γυναίκες γενικότερα, είτε κάποιες ομάδες στόχοι, όπως οι γυναίκες με χαμηλά επαγγελματικά εφόδια, οι υπεύθυνε για τις οικογένειες γυναίκες, για τα παιδιά τους, φαινόμενα γενικά διακρίσεων και φαινόμενα κατά συνέπεια φτώχειας. Η κυρία Μπλινκεβιτσίουτε αναφέρθηκε σε πέντε συγκεκριμένα θέματα περίπλοκα για την κατάσταση των γυναικών. Το πρώτο θέμα έχει σχέση με την νομοθετική κατάσταση που ισχύει σήμερα στην Ευρώπη, την αναθεώρηση δηλαδή της οδηγίας 2006-54 που επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ισότητας ευκαιριών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για να αποφύγουμε διακρίσεις στην απασχόληση. Το δεύτερο θέμα, το οποίο έθεσε η συγγήτρια, είναι η διαφοροποίηση στις αμοιβέ. Το βιώνουμε στην Ευρώπη ακόμα και σήμερα αυτό και υπάρχουν κατηγορίες γυναικών οι οποίες ε, έχουν πολύ εις βάρος τους ε, ε, θα έλεγα αμοιβέ. και αυτό δημιουργεί και προβλήματα και στη σταδιοδρομία και στη συνταξιοδότηση την φτώχεια στις γυναίκες άνω των 60 γιατί δεν είχαν μια πλήρη απασχόληση και γιατί πολύ συχνά ήταν στις χαμηλότερες βαθμίδες των εργαζομένων. Υπάρχει επίσης και το θέμα της εξατομίκευσης των δικαιωμάτων. Υπάρχουν συστήματα που δεν δίδουν τα δικαιώματα αυτά στις γυναίκες, οι οποίες πολύ συχνά σε μια πρώτη φάση σαν απλά Υπάρχει επίσης το θέμα της αγοράς εργασίας, το οποίο συνδέεται με τη διαφοροποίηση των μισθών και των συντάξεων. Εδώ βιώνουμε πολλές διακρίσεις, παθητικές ή ενεργητικές. Στις παθητικές διακρίσεις περιλαμβάνεται και ο συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπου για μια ακόμη φορά οι γυναίκες έχουν τις περισσότερες, τα περισσότερα κοινωνικά βάρη. Γι' αυτό ακριβώς και για το τέταρτο σημείο προτείνεται να τεθεί το θέμα της φτώχειας των παιδιών. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που, που δημιουργείται ανάμεσα στην φτώχεια των οικογενειών, των μητέρων και των παιδιών. Γι' αυτό το λόγο και καλούμε την δημιουργία ενός συστήματος εγγυήσεων για τα παιδιά που θα δίδει δικαιώματα σε επίπεδο δικαίου για να μην εμπλακούν σε αυτό τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Διευκρινίζεται επίσης ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος ρόλος ε, των κοινωνικών εταίρων όπως επίσης και τη σωστή πρακτική σε επίπεδο κώδικα συμπεριφοράς για τις συλλογικέ συμβάσεις, ίση αμοιβή για ίση εργασία και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Άκουσα τις διάφορες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν από τους συναδέλφους και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την προσπάθειά μας για να καταλήξουμε στην πιο δραστήρια λύση για τις γυναίκες. Αν εγκαίρικε, βλέπω δεν ζητάει το λόγο ο Αρναός. Ποιος τελικά. Αν νόμιζα σε να, αλλά όχι. Παρακαλώ, Ευχαριστώ. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε την συντακτή της γνωμοδότησης για τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί πραγματικά είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε με το ζήτημα τη φτώχεια που πλήττει τι γυναίκε, γιατί αποτελεί πραγματικότητα ότι είναι πιο ευάλωτε στον αντίκτυπο τη φτώχεια οι γυναίκε. Ωστόσο, φοβούμαι ότι δεν υπάρχει μια οικονομική ενιαία, οικουμενική συγγνώμη, ενιαία λύση για όλα τα κράτη-μέλη, η οποία θα μπορούσε να εξαλείψει από τη μία μέρα στην άλλη τη φτώχεια. Όμω υπάρχουν κάποιε βασικέ αρχέ, τι οποίε γνωρίζουμε και εάν τηρήσουμε αυτέ τι βασικέ αρχέ, μπορούμε να μειώσουμε τουλάχιστον το επίπεδο της φτώχειας. Το πρώτο από αυτές τις, από αυτά τα, η πρώτη από αυτές τις βασικές αξίες στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ είναι η εκπαίδευση, η παιδεία γενικά. Δηλαδή εάν υπάρχει ένας τρόπος για να ξεφύγει κανείς από την ένδια, είναι ακριβώς ε, το επίπεδο της ε, εκπαίδευσης. Και βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο στην πρωτοβάθμια ή στην δευτερομάθμια εκπαίδευση, αλλά και πέραν αυτής, δηλαδή στη μεταδευτερομάθμια και στην ε, διαβίου κατάρτιση. Μία δεύτερη μέθοδος ή ένα δεύτερος παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να ξεφύγουν από τη φτώχεια είναι ε, το να ε, αποκτούν περαιτέρω δεξιότητες ε, και σε αυτό αναφέρομαι ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα φροντίδα τα παιδιών τα οποία χρήζουν περαιτέρω φροντίδα και υποστήριξη και για παράδειγμα φροντίδα και για ηλικιωμένου. Γιατί πολύ συχνά οι αρμόδιοι για την φροντίδα των παιδιών είναι ηλικιωμένοι ε, οι άτομα με αναπηρία είναι εκείνο τα οποία αναλαμβάνουν την φροντίδα των παιδιών και βέβαια το εισόδημά τους είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οπότε και πάλι έχουμε εδώ το ρόλο της γυναίκας η οποία μένει δηλαδή ε, μόνη της ε, στην οικία με μικρά παιδιά και αναλαμβάνει και αυτό το ρόλο και αντιμετωπίζει και πάλι το πρόβλημα της φτώχειας. Από εκεί και μετά υπάρχει το πρόβλημα ε, των ε, γυναικών που ε, λαμβάνουν σύνταξη, συνταξιοδοτημένες γιατί βέβαια οι αντίστοιχες διαφορές των μισθών υπάρχουν και σε, μεταφράζονται σε αντίστοιχες διαφορές και στις συντάξεις. Δηλαδή βλέπουμε μια διαφορά της τάξης του 23% εδώ σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Ε, πέραν αυτού τώρα υπάρχουν κάποια ε, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν ε, προ όφελο των γυναικών σε κοινωνικά αποκλεισμένε ομάδε. Υπάρχουν μία σειρά από projects τα οποία προσανατολίζονται στην υποστόρευση αυτών των γυναικών, για παράδειγμα microcredits, δηλαδή οι μικροπιστώσεις, ειδικέ κοινοτικού χαρακτήρα δράσεις υποστήριξης στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες με ειδικότερο στόχο τις γυναίκες και από εκεί και μετά θα πρέπει να αναφερθεί ότι ε, οι επιχειρήσεις ε, θα, μπορούν, θα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως ένα εργαλείο για τον να βγουν οι γυναίκες από την φτώχεια. Ευχαριστώ. Λέω πρώτος για να του. Η μάμη Μαριάννα Χάρτιν θα αναλάβει για την άλλη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Λίν για την έκθεση αυτή. Δεν έχω εδώ τις ε, προτάσεις της Γιάννα, μόνο κάποιες δικές μου σημειώσεις, αλλά ξέρω πως ε, έχει σκοπό να συνεργαστεί μαζί σας. Τώρα, από μια γρήγορη ματιά που έριξα, σε αυτή την πραγματικά καλή γνωμοδότηση, στην αρχή αναφερόμαστε στην διαφάνεια στα μισθωτικά συστήματα και υπάρχει και η αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Πιστεύω πως υπάρχει πάντα μια δυσκολία όταν λέμε πως μια γυναίκα και ένας άντρας θα πρέπει να πληρώνονται το ίδιο η εργασία στον ίδιο χώρο και αυτό δεν μπορεί να ισχύσει βέβαια άμα είσαι αποσπασμένο εργαζόμενο. Τώρα τα μισθολογικά λοιπόν κλιμάκια θα πρέπει να είναι απόλυτα διάφανα. Το θέμα βέβαια ξεπερνά αυτή τη διάσταση Εσεί, στην παράγραφο 1 αναφέρεστε σε μια αντιστροφή του βάρους απόδειξη τη της περιπτώσης που καταγγέλλεται διάκριση στον ε, στο χώρο τη εργασία, Διάκριση με γνώμονα το φύλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή πως όλοι είναι αθώοι μέχρι να ε, αποδειχθούν πως είναι ένοχοι. Οπότε ανησυχώ πως οποιαδήποτε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να επηρεάσει όλους τους πολίτες. Δεν θέλω να το διαγράψετε, αλλά πιστεύω πως πρέπει να το συζητήσουμε παραπάνω. Στην παράγραφο 3 αναφέρεστε στις ε, επισφαλείς ε, συμβάσεις. Παρόλο που συμφωνώ πως έχει αυξηθεί ο αριθμός των συμβάσεων τέτοιου είδους, η επισφάλεια δεν έχει να κάνει μόνο με τη διάρκεια απασχόλησης κάποιου εργαζομένου μπορεί να είναι ο τρόπος ε, ε, που πληρώνονται οι ώρες απασχόλησης, ο αριθμός ωρών και τα λοιπά, το κατά πόσο πληρώνονται κοινωνικές εισφορές. Δηλαδή, σκεφτόμαστε ποτέ ε, για αυτή τη βόμβα βραδίας ανάφλεξης όταν κάποια στιγμή τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα βασίζονται στις φορές ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσωρινές συμβάσεις και δεν πληρώνουν κοινωνικές εισφορές. Νομίζω ότι ο χρόνος μετά από τον οποίο θα πρέπει μια τέτοιου είδους ε, σύμβαση να μετατραπεί σε μόνιμη θέση, να σας πω καταρχήν δεν θέλουν όλοι μια μόνιμη ε, θέση εργασίας, αλλά ίσως εδώ θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση η οποία θα διευκολύνει του να δίδονται τέτοιου είδους συμβάσεις ε, χωρίς να συμπεριλάβουμε φρασιολογία τόσο επιτακτική όπως αυτό το πρέπει, το must. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται εδώ που είναι η καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ε, ένα θέμα στο οποίο είχαμε πολλές επιτυχίες στην Ιρλανδία όπου επιδοτήσαμε όχι τους παιδικούς σταθμούς αλλά την ε, καλύτερη εκπαίδευση για παράδειγμα των όσων εργάζονται σε αυτούς των πιογωγών, των βρεφοκόμων κτλ. Πρέπει δηλαδή η διατύπωση που επιλέγουμε να μην κάνει διάκριση εναντίον των ε, γυναικών που αποφασίζουν να μείνουν οι ίδιες στο σπίτι να φροντίσουν την οικογένειά τους. Ίσως λείπει αυτή η λέξη από εδώ, δεν ξέρω αυτά τα 80 εκατομμύρια ανθρώπων που βοηθάνε στο σπίτι, εντάξει, οι περισσότερες από αυτές είναι γυναίκες. Υπάρχει και, υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι εργάζονται στον κλάδο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως γυναίκες, οπότε καλό είναι να μείνει. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση στην πέμπτη παράγραφο είναι αυτή, αυτό το συνταγματικό δικαίωμα σε άδεια με αποδοχές ε, σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Και είπα, γιατί να το περιορίσουμε σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αν λειτουργεί αλλού, θα έπρεπε να δούμε τι ακριβώς κάνουν στην Αυστραλία και αλλού και ίσως να εφαρμόσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Και τέλος, συμφωνώ μετά όσα ακούστηκαν για ε, τις γυναίκες επιχειρηματίες, για την μικροχρηματοδότηση. Έχουμε τέτοια σχέδια κειμένων στην Επιτροπή μας και όλα αυτά τα μικρά μικρά κομματάκια θα συνθέσουν αυτό το πάζλ που θα καταπολεμήσει τη φτώχεια που ε, εξαρτάται από το φύλλο. Οι γυναίκες ξέρετε πως είναι ε, η μεγαλύτερη ομάδα ε, που λαμβάνει μικροδάνεια ή μικροχρηματοδότηση. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας πω πως η συνάδελφος Γιάννα πραγματικά λυπάται που δεν μπορούσε να παραβρεθεί σήμερα. Thank you, Chair. Um, I'm uh, representing my colleague. Η κυρία Ράντια για τους πράσινους. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Εγώ Ευχαριστώ την συνάδελφο Μόνικα. Από την ε, πλευρά μας και εμείς να πούμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το σχέδιο και αναμένουμε βέβαια με ε, ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις ε, που θα γίνουν θα πρέπει εμείς ε, κατά τη δική μας άποψη να εστιάσουμε σε τέσσερα ε, σημεία. Κάποια ε, βέβαια ήδη αναφέρονται τμήματικά μέσα στο σχέδιο, αλλά θα θέλαμε να τονιστούμε περισσότερο καταρχήν σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επισφαλούς απασχόλησης και των μισθολογικών διαφορών, γιατί βλέπουμε συχνά να πέφτουν σε ένα είδος παγίδας οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, δηλαδή συχνά είναι αναγκασμένες να δουλεύουν όχι σε καθεστώ πλήρου απασχόληση, αλλά μερική απασχόληση. Εμεί θέλουμε λοιπόν να ε, μπορούν να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να μην ε, βρίσκονται σε επισφαλή, επισφαλή απασχόληση. Και βέβαια, ε, ειδικότερα η φτώχεια που αφορά του ηλικιωμένου έχει γυναικείο προσφύλλο. Δηλαδή, είναι περισσότερε οι γυναίκε οι οποίε πλήττονται από αυτό το είδο φτώχεια. Οπότε θέλουμε να έχουμε περισσότερε γυναίκε οι οποίε έχουν πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια τη ε, ζωής τους ως οικονομικά ενέργειες. Από εκεί και μετά ε, ένα ακόμα ε, Ε, σημείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αν ε, δούμε το φορολογικό σύστημα σε διάφορα κράτη-μέλη θα δούμε ότι υπάρχει ακόμα ε, μία διακριτική μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων άρα θα πρέπει να αναφέρεται αυτό γιατί πραγματικά έχει επιπτώσεις στον ρολογινετών μέσα στην κοινωνία οπότε να πρέπει να γίνουν κάποιες εδώ πρόοδοι και να αυξηθεί βέβαια και αυξηθούν οι σχετικέ δαπάνε σε κρατικό επίπεδο για αντίστοιχε επενδύσει όπω για παράδειγμα ε, υποδομέ φροντίδα ε, παιδιών αλλά και άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ ε, και αυτό είναι και το τρίτο από τα σημεία που θα θέλαμε να αναφέρετε. Θα πρέπει δηλαδή ειδικότερα οι επενδύσει σε κοινωνικέ υπηρεσίε να αυξηθούν όπω για παράδειγμα η λήψη υπόψη στο πλαίσιο των προπολογισμών της διάστασης ε, του φύλου, αυτό το gender budgeting δηλαδή, ούτως ώστε να είναι ε, καλύτερη η κατανομή των ε, σχετικών δαπανών μεταξύ των δύο φύλων. Και ένα ακόμα σημείο τέλος το οποίο έχει αναφερθεί αλλά συχνά δεν λαμβάνει την έμφαση που πρέπει είναι ότι όταν ε, ε, οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με την φτώχεια. Έχουμε να κάνουμε κυρίως ε, με μετανάστες και πρόσφυγες, γυναίκες οι οποίες απλούνται οπότε θα πρέπει να αναφέρονται. Αναφέρεται και αυτή η διάσταση. Αυτές λοιπόν, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά ζητήματα και η Μόνικα Βάνα, δική μας δηλαδή στη Όδηση Συγγήτρια θα συμμετάσχει με μεγάλο ενδιαφέρον σε ειδικέ συζητήσει που θα γίνουν με του υπόλοιπου σκιώδη συγγητέ και την ίδια την συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ε, Μάρα Πιτσότου για την, για e Oui, euh, Monsieur le Président. Je remercie Madame Boylan pour son rapport. Euh, euh, Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Προοπτικές από πλευρά των φίλων. Ε, θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε λοιπόν πώς να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γυναικών. Εδώ δεν ε, έχω αμφιβολίες για την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται, αλλά παρόλα αυτά στο σημείο 4 λέει ότι η φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να έχει αντιμετωπίσιμο κόστος. Πώς αυτές οι αντιμετωπίσιμου κόστου υπηρεσίες για τα παιδιά έχουν σχέση με τον μισθό των γυναικών που εργάζονται. Στο σημείο 5, ε, η οικιακή βία στις φτωχές γυναίκες είναι θέμα, αλλά τι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε γιατί υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν μορφές βίας εις βάρος των γυναικών και στις, ε, στις πλούσιες οικογένειες. Όλο και πιο πολλές γυναίκες στήγονται από αυτό. Και αυτές οι, οι μορφές βίας υπάρχουν στους λεγόμενους νεοεισερχόμενους πληθυσμούς. Ταυτόχρονα ε, διάκριση ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπω τον τρόπο μέσω της αύξησης του μισθού των γυναικών που έχουν προσωρινές θέσεις απασχόλησης, ε, πώς αυτό θα μειώσει την ανεργία και θα ενισχύσει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Μου φαίνεται λίγο άσχετο. Για το σημείο 3. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όλα λέγονται εδώ, στο σημείο 3. Ότι η συγκέντρωση των γυναικών σε προσωρινές θέσεις απασχόλησης είναι δυσανάλογη και μη θελημένη. Δυσανάλογη και συχνά μη θελημένη, Αυτό σημαίνει ότι είναι καταδικασμένες οι γυναίκες, ότι δεν πηγαίνουν να πάρουν τη θέση αυτή εργασίας γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δουλεία εις βάρος των γυναικών. Και η λύση δεν είναι εδώ, σας το έχω ήδη πει. Το είπε ο εισηγητής, αλλά δεν το έχει γράψει. Μήπως θα μπορούσαμε να αφήσουμε τις γυναίκες ελεύθερες να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και όχι να τις καταδικάζουμε σε προσωρινές θέσεις απασχόλησης και νομίζω ότι η λύση περνάει από τον οικογενειακό μισθό μαθητείας, είτε για τον πατέρα είτε για τη μητέρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο οποίος ωφελείται από το συγκεκριμένο μέτρο είναι αυτός ο οποίος έχει τη χαμηλότερη αμοιβή. Αυτή είναι η άποψή μας. Νομίζω ότι το σημείο 3 είναι ενδιαφέρον αλλά το υπόλοιπο ψήφισμα είναι λιγάκι άσχετο με το θέμα. Τελευταία λοιπόν παρέμβαση, οπότε θα δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μανουέλα Αγγελέν και η Ευελίνα, Ευελίνα Άστο. Βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, θα πάρει το λόγο αν θα μοιραστείτε το χρόνο σας. Ε, αναφέρθηκε δικαίως ότι ε, οι χαμηλότεροι μισθοί για τις γυναίκες ε, τελικά έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερο ότι ψηλότερη φτώχεια για τι γυναίκε και πράγματι ο κίνδυνο ε, να υπομένουν τη φτώχεια οι γυναίκε είναι υψηλότερο σε μεγαλύτερε ηλικίε. Η Επιτροπή έχει εστιάσει τι δικέ τη εργασίε ε, σε μέτρα τα οποία μπορούν ακριβώ να αντιμετωπίσουν αυτού του ε, παραγόντε οι οποίοι δεν επιτρέπουν στι γυναίκε να συμμετέχουν και στην αγορά εργασία. Και στο, στη, στο λευκό paper σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, συνταξιοδότηση των γενικών, αναφέρεται αυτό το ζήτημα, αλλά και άλλο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα ειδικότερα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία ε, τονίζουν και έχουν τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη του να ε, παρέχεται ε, ε, κατάλληλη και οικονομική βέβαια φροντίδα των παιδιών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο για τα κατάλληλα κίνητρα για την απασχόληση. Αναφέρθηκε επίσης εκεί και η μείωση της μισθολογική διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Τώρα σε ό,τι αφορά τον εγγύηση για το child guarantee, να πούμε ότι ήδη υπάρχει εδώ σε ε, ε, ένα εργαλείο σε ό,τι αφορά ε, τις επενδύσεις και τα διαφθορτικά ταμεία ειδικότερα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προβλέπει τέτοιου είδους project, δηλαδή σε ό,τι αφορά υψηλή ποιότητα υπηρεσίας φροντίδας παιδιών, αλλά και υποδομές για την φροντίδα των παιδιών και υποδομές για την εκπαίδευση των παιδιών. Επίσης, προβλέπονται εδώ ειδικέ δομέ για την υποστήριξη τη ε, ασφαλού ε, ε, των οικογενειών και τη υποστήριξη τη περαιτέρω. Μία περαιτέρω πρωτοβουλία για την υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου στοχεύει στην ακριβώς την πιο δίκαια κατανομή των σχετικών μεταξύ των δύο φύλων και κατά συνέπεια θεωρούμε πως και αυτό το μέτρο μπορεί με τη σειρά του έμεσα αν θέλετε να έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών μέσω δηλαδή αυξημένης ε, συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μείωση της αντίστοιχης ε, φτώχειας ε, των γυναικών. Τέλος να πούμε ότι συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά μια έκθεση που θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την φτώχεια των δύο φύλων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εκδοθεί μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2016. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της σήμερα σας διάταξης. 28 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών και 16 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 15 της σημερινής σας διάταξης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ειδικότερα ε, τις ε, οικονομικές και ε, κοινωνικές πτυχές η συγκήτρια είναι Σοφία Ριμπέρου οπότε της δίνω το λόγο για να περάσουμε σε συζήτηση των τροπολογιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την περασμένη Δευτέρα λάβαμε 430 τροπολογίες από το σύνολο των πολιτικών ομάδων, οπότε αυτό δείχνει τη μεγάλη δέσμευση, του υψηλό βαθμό δηλαδή ενδιαφέροντος ε, που υπάρχει από την πλευρά όλων ε, των προβουλευτών ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές με όλες τις προτάσεις οι οποίες έγιναν σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, προκειμένου δηλαδή να επικεντρώσουμε καλύτερα στις δράσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κοινωνικά ζητήματα. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιε πρώτε προτάσει με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Ε, μέχρι στιγμή οι διαπραγματεύσει που έχουν γίνει ε, ε, έχουν ακολουθήσει μια καλή ε, πορεία. Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει ελπίδα <laughs> να υπάρξει ένα συνενετικό κείμενο. Έχουμε καταλήξει σε συνολικά 54 συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες αντιστοιχούν σε 264 αρχικές τροπολογίες οπότε εδώ και τρεις-τέσσερις εβδομάδες ουσιαστικά μετά από την ε, υποβολή των ε, τροπολογιών. Θα έχουμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις εβδομάδες, μετά έχουμε και μια εβδομάδα ε, μια την πράσινη εβδομάδα και την εβδομάδα του, της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για μας, τα οποία θα πρέπει να ε, συζητηθούν λεπτομεριακά και ήδη έχουν ε, συζητηθεί για παράδειγμα οι συντάξει, το flexicurity, το επανομαζόμενο, τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι κοινωνικέ συνθήκε εργασία και ούτω καθεξής. Όμω ε, σε κάθε περίπτωση εδώ θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα ικανοποιεί όλε τι πολιτικέ ομάδε και θα έχουμε ταυτόχρονα ένα δυνατό κείμενο το οποίο θα εκπροσωπεί σωστά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ με αυτή την παρέμβαση θα ήθελα να πω ότι είμαι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το στόχο να δώσουμε δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη κοινωνική διάσταση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και γι' αυτό είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ με όλε τι ε, πολιτικέ ομάδε, δηλαδή μέσω των σκιώδων συζητητού του, για να το επιτύχουμε ε, και να του ευχαριστήσω ήδη για την ε, πολύ μεγάλη ειλικρίνεια που επέδειξαν ήδη κατά τι προκαταρκτικέ μα εργασίε. Ευχαριστώ. Ήσασταν σύντομοι και περιεκτικοί Σέντζο ε, Κουτιέρες έχει το λόγο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη Σοφία για τη δουλειά που έκανε και για το γεγονός πως ε, είναι τόσο δεσμευμένη που σε χρόνο ρεκόρ και με τέτοιο αριθμό τροπολογιών έχει ξεκινήσει ε, με αυτή τη δουλειά. Οι τροπολογίες των σοσιαλιστών θέλουν να καλύψουν τρία ουσιαστικά θέματα, την απασχόληση, τη μάχη κατά των ανισοτήτων και την ε, διακυβέρνηση της Ευρώπης, την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Εμείς θεωρούμε πως την απασχόληση θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για κάποια θέματα. Καταρχήν, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε ούτε με τον αριθμό ε, θέσεων εργασίων, εργασίες που δημιουργούνται, ούτε με την ποιότητα αυτών κατανοούμε πως ε, σε μεγάλο βαθμό οι εργασιακές ε, αναθεωρήσεις που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία εις βάρος της ασφάλειας και μια διαφορετική κατανομή των ε, θέσεων εργασίας χωρίς να έχει αυξηθεί η ωριά παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουν μειώσει για παράδειγμα ε, τις ώρες εργασίας, ε, δίνουν ε, συμβάσεις ωριές και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε βελτίωση ούτε ποιοτική εργασία. Θέλουμε λοιπόν μία, αν θέλετε, επικριτική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει, γιατί οι διαστοδετικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν ε, με μία αξιολόγηση αυτών που εισήχθησαν στο παρελθόν και με μία βελτίωση ή αλλαγή ε, κάποιων διατάξεων έτσι ώστε να υπάρχει μία ίση σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ευελιξίας αυτής που είναι απαραίτητη. Θα πρέπει λοιπόν την νομοθεσία να την προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες, αλλά να είναι προστατευτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο Σαββατοκύριακο μας είπε πως είμαστε ευάλωτοι και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η ανάπτυξη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ε, ευάλωτη λόγω τιμής πετρελαίου, λόγω ε, αναπτυσσόμενων χωρών, ε, ίσως επειδή δεν χρησιμοποιούμε τον σωστό τρόπο το σχέδιο Juncker, είτε γιατί υπάρχουν κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή τις προγραμματισμένες επενδύσεις για να χρησιμοποιήσουν το πακέτο Juncker. Άρα λοιπόν έχουμε μία μείωση των επενδύσεων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο κάνει πολύ ευάλωτη την ανάπτυξή μας και θα πρέπει για μια φορά ακόμα να προσπαθήσουμε οι επενδύσεις σε εμάς να μην εξαρτώνται από την οικονομική συγκυρία τρίτων χωρών, να ενισχύσουμε τη θέση μας. Και το τρίτο είναι η μάχη κατά των ανισοτήτων που είναι ένα πρόβλημα μακροοικονομικό και κοινωνικό ε, που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψαλίδα μεταξύ αυτών των εχόντων και των μη εχόντων, ε, που δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες γιατί υπάρχουν ε, ομάδες που πλήττονται και η ψαλίδα μεγαλώνει συνέχεια πρώτα απ' όλα λόγω της άδικης φορολόγησης και λόγω της καταστροφής ή εν πάση περιπτώσει ε, μειωμένης ε, στήριξης του κοινωνικού ε, συστήματος που έχουν, του συστήματος κοινωνικής προστασίας και παράδειγμα με το συνταξιδοτικό, με τα επιδόματα αναργίας, τα οποία μειώνουν αυτό το επίπεδο προστασίας που ήταν κάτι το οποίο εξασφάλιζε την κοινωνική συνοχή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Pilar de nuestras enmiendas es que cuando hablamos όταν μιλάμε λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο για διαρθρωτικές αλλαγές, εκτός από το ότι θα πρέπει αυτό να το μεταφράσουμε, γιατί εντάξει είναι ένα μάντρα το οποίο τα καλύπτει όλα, οπότε εμείς θα πρέπει να δούμε τι είδους μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε, γιατί πολλές είναι ε, στα σκαριά, η βασική είναι η διακυβέρνηση του ευρώ. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για πρώτη φορά να έχουμε μία σύσταση συγκεκριμένη που θα απευθύνεται στις χώρες του ευρώ και να τη χρησιμοποιήσουμε για να πούμε πως χρειάζεται μια οικονομική διακυβέρνηση του χώρου του ευρώ. Εμείς μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, ελάχιστου μισθού, ένα διευρυμένο πλαίσιο με μια γκάμα μισθών, έτσι ώστε να μην έχουμε εργασιακή φτώχεια, να μην έχουμε μισθούς που είναι κάτω από το επίπεδο που επιτρέπει να ζήσει με αξιοπρέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε με το τι θα γίνει με τους αυτόματους σταθεροποιητές στην απασχόληση στην Ευρώπη, όλα αυτά είναι προτεραιότητες για την ομάδα μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι τροπολογίες οι οποίες περιγράφουν τη θέση μας και είμαστε έτοιμοι και διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό και να είναι μια γνωμοδότηση την οποία θα στηρίξει όλη η Επιτροπή μας. Ο Άννα λοιπόν θα μιλήσει εξ ονόματός της. Ναι. Εκ μέρους λοιπόν της αστείωσης της ηγετρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ριμπέρου, την εισηγήτρια, για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τους συμβασμούς η σκιώδη συγκήτρια μας ε, υπέβαλε 25 ε, τροπολογίες οι οποίες ήδη έχουν ε, ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται για τις εμβαστικές τροπολογίες και ήδη εμείς έχουμε από δική μας πλευρά αποστείλει τις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά τις εμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ πιο συγκεκριμένα ένα-δύο σημείο. Καταρχήν, συμφωνούμε με τη γενικότερη κατεύθυνση που ακολουθεί το κείμενο και ε, με τις τροπολογίες. Δηλαδή οι δικές μας τροπολογίες από δική μας πολιτική ομάδα έχουν αναφερθεί στα ζητήματα της ε, επικουρικότητας και της των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατομελών αλλά και ε, σε ό,τι αφορά τις διαφορές μεταξύ των κρατομελών, των διαφορετικών επιπέδων απασχόληση και των διαφορετικών τύπων των αγορών εργασία. Αναφερθήκαμε επίση και ε, στον ρόλο που μπορεί να παίξει εδώ ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αναφερθήκαμε σε μια ε, ε, σειρά από προβλήματα τα οποία θεωρούσαμε πως υπήρχαν στις συμβαστικές τοπολογίες που κυκλοφορήσει μέχρι τώρα και συντακτικού χαρακτήρα. Θα υπάρξει βέβαια αύριο το πρωί μία ακόμα συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, οπότε θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο σε εκείνη τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, το Πρόεδρος. Ο Λάτωνα. Ε, θα μιλήσετε εσείς ή κάποιος άλλος για την άλλη, όχι. Εγκάβιτ σήμερα, λοιπόν, για την Κούα. Ευχαριστώ πολύ. Ως Γκούα, εμείς από την δική μας πλευρά. Θέλουμε η έκθεση, η ετήσια έκθεση ανάπτυξη συναλάβει υπόψη και διάφορα ζητήματα που οποία συζητήσαμε και προηγουμένως, δηλαδή ότι ε, το ε, Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν του ώστε κάποια στιγμή να επιτύχουμε το τριπλό αυτό α στο κοινωνικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα οποία αναφέρονται στην έκθεση μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν καταδεικνύουν ότι θέλουμε να δώσουμε ή θέλουμε να συμβάλλουμε, ε, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ε, σε μια αλλαγή της κατεύθυνσης, της κακής κατεύθυνσης που ακολουθούμε μέχρι τώρα. Ε, εμείς έχουμε βάλει 18 τροπολογίες, να μείνουμε κάτω από το ψυχολογικό όριο, αν θέλετε, των 20. Ε, σε κάποια δηλαδή, σήμερα αποφασίσαμε να απόσχουμε, αλλά κάναμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες ακολουθούν την γενική κατεύθυνση ως εξής. Με την ετήσια έκθεση ανάπτυξης βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένα επίπεδα επισφαλούς απασχόλησης, φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας και αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η έκθεση θα πρέπει να ε, ασχοληθεί και με ζητήματα τα οποία ε, σχετίζονται για παράδειγμα με το νέο κάλεσμα που ακούμε για την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασία, στο Flex Security, που μπορούμε δηλαδή να οδηγήσουμε τη σειρά στην αύξηση της επισφολής απασχόλησης. Εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε ξεπεράσει αν θέλετε το Flex Security, αλλά βλέπουμε τώρα ότι τίθεται και πάλι νέες προτάσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίες νέες επενδύσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην ε, ε, κοινωνική ε, πολιτική, δηλαδή διασφάλιση των θέσεων εργασίας, για ε, της λιτότητας, ε, διασφάλιση ελάχιστων εισοδημάτων, ελάχιστων, ελάχιστων συντάξεων ε, και ακριβώς αυτή τη γενική κατεύθυνση ακολουθούμε τροπολογία μας. Για παράδειγμα, η τροπολογία 43 σε ό,τι αφορά την νεοτολογική σκέψη α, να πούμε ότι ναι, σταδιακά έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σε απαράδεκτα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν καλό είναι να το κάνουμε δηλαδή να ε, ασκήσουμε κριτική και σε διαφορετικές αλλαγές, ε, διαφορετικές ε, μεταβολές ή μεταρρυθμίσεις οι οποίες μειώνουν τα δικαιώματα για παράδειγμα των εργαζομένων. το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί και η τροπολογία μας σε ό,τι αφορά την σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία. Δηλαδή, κατά δική μας άποψη, ναι, ε, πολλά άτομα δεν ε, λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατά συνέπεια δεν βρίσκουν πρόσβαση στην αγορά εργασία, αλλά από την άλλη πλευρά οι διάφορε περικοπέ των ε, κατοικών προπολογισμών που έχουν λάβει η χώρα σε διάφορα κράτη-μέλη έπλεξαν ειδικότερα το τομέα τη επενδύα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Μετά, σε ό,τι αφορά στη συμβαστική τοπολογία για τον αιτιολογή ε, και πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, με το ζήτημα της μη ε, τυπικής μη επίσημης εκπαίδευσης και το ε, πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει ή όχι τις δυνατότητες απασχόλησης. Θα πρέπει να αναφέρεται λοιπόν αυτό το ζήτημα με περισσότερη έμφαση από ό,τι γίνεται τώρα και μετά σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τοπολογία F να πούμε ότι γίνεται στο κείμενο, μία αναφορά στην, ε, στα επίπεδα της Τόγιας κατά, τις ε, τελευταία, έτη, στο πλαίσιο και των στατικών στόχων της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα λοιπόν συμβαστική τροπολογία αναφέρεται ότι τα επίπεδα της φτώχειας έχουν σταθεροποιηθεί κατά τα έτη 2013-2014. Εγώ θα ήθελα ε, να ακούσα από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία, ποια είναι η πηγή τους, γιατί τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τον Eurostat δεν τα έχουμε λάβει ακόμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας έλεγχος προτού συμπεριληφθεί αυτό το, μια τέτοια αναφορά ε, ε, ε, σε, μια, σε ένα τέτοιο κείμενο. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε λόγο για μια εντύπωση που έχουμε η οποία τελικά όμως δεν είναι επιβεβαιωμένη στα κράτη-μέλη. Μετά σε ό,τι αφορά την παράγραφο 13, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον εξυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο βασίζεται στην ζήτηση να πούμε ότι εμείς λυπούμεθα για το γεγονό ότι εδώ ουσιαστικά δεν έχουμε επιτυχεί πρόοδο, το αντίθετο έχουμε κάνουμε κάποια βήματα προ τα πίσω. Και εδώ σα υπενθυμίζω και το έτο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σα αναφέρω ότι όταν κάνουμε λόγο για τον εξυγχρονισμό ε, των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μα και τι επιπτώσει που έχουν στην υγεία συγκεκριμένα τύποι επαγγελμάτων. Ε, άλλοι παράγοντε, για παράδειγμα, είναι ε, η γύραση του πληθυσμού, το προσδόκιμο ε, της ζωής και το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουμε ε, τους κατάλληλους μισθούς λαμβάνοντας υπόψη και το σύγχρονο φαινόμενο της μετανάστευσης. Έχουμε υποβάλει τη δική μας τροπολογία σε ό,τι αφορά την παραγραφό 14 που βρίσκεται το κατάλληλο, την κατάλληλη ισορροπία και από εκεί και μετά δύο ακόμα σχόλια θα ήθελα να κάνω σε ό,τι αφορά δύο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί εδώ ε, στις δικές μας τροπολογίες, δηλαδή το ένα αφορά τους άστεγους ανθρώπους και από εκεί και μετά το δεύτερο αφορά τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι υπηρεσίες ε, για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού ε, να γίνεται λοιπόν λόγος ότι χρειαζόμαστε έναν υγιή ανταγωνισμό ο οποίος θα αναδεικνύει τα καλύτερα και όχι απλά τα φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά από την πλευρά μας ως προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε περισσότερο την αλόγω έκθεση. Η Τζιν Lambert τώρα για τους ε, πράσινους. Θα συμφωνήσω και εγώ με αυτούς οι οποίοι εκφράστηκαν θετικά για την ε, εισήγηση. Αποτελεί πράγματι μια καλή βάση για συζήτηση. Καταθέσαμε πολλές τροπολογίες δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, μάλλον κάποιες από αυτές περνούν σε λεπτομέρειες, κάποιες άλλες είναι κατευθυντήριες θα έλεγα, που βελτιώνουν την ποιότητα της δουλειάς την οποία κάνουμε. Ένα από τα πράγματα στα οποία θέλουμε να πιέσουμε κάπως περισσότερο είναι η διάσταση καταπολέμησης της φτώχειας. Τι προσπαθούμε ακριβώς να κάνουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί επανειλημμένα για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Τα συστήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Και φυσικά οι μισθοί παίζουν εδώ τον καθοριστικό ρόλο, υποτίθεται. Καταφέσαμε λοιπόν πολλές τροπολογίες και για το θέμα της κατοικίας αντίστοιχα είναι κομβικό και περιλαμβάνεται σε πολλές ε, συστάσεις σε διάφορα σημεία για κάποια κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν υπάρχει κατοικία με σωστό τρόπο αυτό έχει επιπτώσεις και σε επίπεδο απασχόλησης και σε επίπεδο υγείας κτλ. βλέποντας την κατάσταση της κατοικίας σε ορισμένες χώρες. Καταθέσαμε επίσης και τροπολογίες για την περιβαλλοντική διάσταση. Γιατί εμείς θέλουμε να τονίσουμε την κατεύθυνση μιας οικονομίας η οποία μειώνει τη χρήση των ορυκτών καυσίμων όλο και περισσότερο και στα πλαίσια της διαδικασίας του εξαμήνου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε με τον εισηγητή τις τροπολογίες νομίζω ότι αποτελούν μια καλή βάση για τις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς ένα τόσο μεγάλο αριθμό τροπολογιών, αλλά είναι καλό να ξεκινήσουμε όσο νωρίτερα γίνεται. Και εγώ κάθε πρωί δίνω μάχη σε ό,τι αφορά το work-life balance μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Ριμπέιρο, η οποία έλαβε εν πολύ υπόψη τις δικές μας θέσεις μέσω των τροπολογιών που καταθέσαμε. νομίζω ότι δεν καταθέσαμε πάρα πολλέ και ελπίζουμε και είναι χαρά μας το ότι είδαμε ότι ελήφθησαν υπόψη. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα βέβαια στην έκθεση αυτή όταν μιλάμε για τις διαφθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για τις διαφθρωτικές αλλαγές, Είναι βασικό να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να δούμε ακριβώς ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχουν ε, προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές ε, ε, εκεί που έχουν επιβληθεί. Δεν μιλάμε πια για την Ελλάδα και αυτό είναι καλό, αλλά έχουμε θα έλεγα κάποια ξεκάθαρα παραδείγματα για τις προσπάθειες επιδίωξης μιας κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία δυστυχώς οδηγεί στο ναυάγιο του Τιτανικού. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν η συνάδελφος να λάβει υπόψη και κάποιες περισσότερες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις τις οποίες οι μεταρρυθμίσεις οι διαφορετικές μπορεί να έχουν σε επίπεδο και κοινωνικό και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρξει μία από κοντά παρακολούθηση για το πώς εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα μέτρα και πώς γίνονται πραγματικότητα, γιατί πάρα πολύ συχνά δυστυχώς και αυτό είναι ένα από τα, ένας από τους περιορισμούς που έχουμε, είναι ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις πραγματικές επιπτώσεις. Η Ευρώπη προσπαθεί να είναι ενημερωμένη για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, αλλά θα πρέπει και σε εθνικό επίπεδο ε, να γίνεται μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων ιδιαίτερα στην φάση όπου ζητείται από την αγορά εργασίας μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά όχι περισσότερη κοινωνική προστασία. Είμαι λοιπόν περίεργη και θα ήθελα να ξέρω πώς ο Υπουργός κύριος Παντοάν αύριο θα έρθει να μας μιλήσει. Θα έρθει εδώ να παρουσιάσει τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα αυτά. Υπάρχουν τέτοιες εγγυήσει σε διάφορες χώρες, αλλά όχι στην Ιταλία. Εκεί έπρεπε να θέσει το ερώτημα λοιπόν. Έχει σημασία με λίγα λόγια το πώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Ένα άλλο θέμα είναι οι συντάξει και οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον τομέα των συντάξεων, του πυλώνα του συνταξιοδοτικού. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με δύο θα έλεγα όψεις. Από τη μία, ε, βλέπουμε την ανάγκη που υπάρχει για την ε, διεύρυνση της εργασιακής ζωής. Από την άλλη δεν έχουμε τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αντιφατικό. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά πάλι τις συντάξεις. Η δημοσιονομική πίεση η οποία θα έλεγα επηρεάζει αρνητικά μέσω της φορολογίας και της επιχειρήσης εμποδίζει την δημιουργία των θέσεων εργασίας. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια κάποια προσπάθεια έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας να μπορέσει να, να... φανεί ε, ευέλικτος εκεί όπου υπάρχουν ε, ελλείψεις. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και εναλλακτικέ λύσεις για αυτούς οι οποίοι δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης ε, Υπάρχουν πολλά κρίσιμα σημεία τα οποία αφορούν και τη συνταξιοδότηση. Η συνάδελφος ίσως θα μας κάνει κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Και ταυτόχρονα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία, η φτώχεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή τις χώρες έχει αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στις διαδικασίες της εκπαιδευτικές των παιδιών Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε τις διαδικασίες αυτές εκεί όπου οι οικονομικές συνθήκες και η οικονομική συντηρία δεν το επιτρέπει. Ε, είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια, το πεδίο άλλωστε προσφέρεται πάρα πολύ. Μάρα λοιπόν, την οποία όμως δεν βλέπω εδώ μαζί μας, οπότε θα δώσω λόγο στην Επιτροπή ο κύριος Ζωρέν κυρία ε, Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Έχουμε παρακολουθήσει την ε, συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε και την ε, γνωμοδότηση. Πολύ ωραία που σας θα δώσω σύντομος. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος που να έχει δει στο λόγο. Οπότε θεωρώ πως έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης. Ναι, δεν έδωσα το λόγο στην εισηγήτρια, βλέπω πως το ζητάει παρόλα αυτά, οπότε παρακαλώ, έχει το λόγο κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα βέβαια με πολύ προσοχή τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι και ε, έκαναν τις σημειώσεις μου. Απλά σα υπενθυμίζω ότι αύριο στι 8 το πρωί έχουμε μια συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Οπότε ε, α προσπαθήσουμε εδώ να είμαστε συνεπεί σε ό,τι αφορά ακριβώ την ισορροπία μεταξύ τη οικογενειακή και τη επαγγελματική μα ζωή. Τώρα, ε, θα ήθελα απλά να δώσω ε, ένα γενικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά την βαστή κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Η κυρία Τσίμερ που αναφέρθηκε στους δείκτες της φτώχεια, να πούμε η Ούλα Τόρνε, ε, που είναι αντιπρόεδρος αυτής εδώ της Επιτροπής με την τροπολογία 91 ε, που έκανε έχει ε, καταφέρει να μπουν αυτοί οι δείκτε για τα δύο τελευταία έτη, 13 και 14 και μετά από εκεί και μετά. Σε ό,τι αφορά το flex security αναφερόμαστε ακριβώς ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο διαστάσει, δηλαδή ναι μεν ευελιξία, απαραίτητη ευελιξία για τι επιχειρήσει, αλλά από την άλλη πλευρά ασφάλεια, δηλαδή διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ούτω καθεξή. Σε καμία περίπτωση εμεί δεν προσπαθούμε εμεί να διασφαλίσουμε τον επιβληθεί αν θέλετε περισσότερο ευελιξία στην, ε, στην ασφάλεια. Προσπαθούμε να τονίσουμε ε, το, την, τη σημασία που έχουν και, ε, και οι δύο πυλώνες αυτοί. Από εκεί και μετά. Όταν αναφερόμαστε στην εποχιακή εργασία ή στην επισφαλή εργασία γενικά, θα πρέπει να μην δώσουμε την ενθασμένη εντύπωση. Εκείνο που αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για μας ως Επιτροπή είναι να αναφέρουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ταξινομήσουμε ή να διαχωρίσουμε την εργασία η οποία πραγματικά είναι απαραίτητη με αυτή τη μορφή και την εργασία εκείνη η οποία αποτελεί εκμετάλλευση των ε, εργαζομένων. Τώρα, ε, ε, σε ό,τι αφορά τους στόχους του οποίου θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο στόχοι σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Καταρχήν θα πρέπει να είναι πολύ καλά στοχευμένες σχετικές επενδύσεις ώστε να δημιουργούν Περισσότερε ακόμα επενδύσει. Δεν θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια λογική απλά ενισχύσεων, ενισχύσεων προς τα κράτη-μέλη. Όχι, θα πρέπει να δίνει τι κατάλληλε δυνατότητε στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τι επενδύσει του η υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνική διάσταση η οποία θα έχει αντίκτυπο, πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Άρα λοιπόν όταν κάνουμε λόγο για ε, κοινωνική προστασία των πολιτών, ακριβώ κάνουμε λόγο ε, για αυτέ τι κοινωνικέ μεταρρυθμίσεις οι οποίε θα πρέπει, διαθωτικέ μεταρρυθμίσεις, οι οποίε θα επιτρέψουν ακριβώ ε, την προστασία των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι εποφελούνται λιγότερα από τα σχετικά δικαιώματα ε, και ακριβώ αυτό είναι και το νόημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να λάβουμε υπόψη μα ε, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε με τρόπο διαφοροποιημένο στι εκάστοτε ανάγκε του, ώστε να του δώσουμε τη δυνατότητα ένταξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι λοιπόν, αυτά είναι ήδη διακήρυξη των βασικών αρχών που διέπουν αυτό το σχέδιο και από εκεί και μετά βέβαια αύριο το πρωί θα έχουμε, όπως είπαμε, την συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών να συζητήσουμε αυτά τα θέματα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν κάνετε, κυρία Ριμπέρο, μια εισαγωγή στην αυριανή συζήτηση ε, των εισηγητών, εισηγητών. Καλώς, ε, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Για τα 17 λοιπόν Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε ε, από αυτού του σχεδίου νομοδότησης. Ε, να σας υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά από τις αύριο στι 2 στις 3 ε, έχουμε την ανοιχτή συνεδρίαση των ε, συντονιστών με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλιση κατά της ανεργίας. Οπότε σας καλώ να παρεμπληθείτε όλοι εδώ. Εμείς θα συνεδριάσουμε στις 17 Φεβρουαρίου από τις 9 ως τις 12 και από τις 3 έως τις 6.30 και μετά την επόμενη μέρα από τις 9 ως τις 12. Αυτά έχω εδώ καταγεγραμμένα. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε σήμερα και καλό σας βράδυ.